Uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το τελευταίο μέρος της ε, συνεδρίασής μας της Επιτροπής Ήτρε. Μέχρι τις 6 θα διαρκέσει η συνεδρίασή μας. Πάμε στο σημείο 14, την Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Πληροφορικής Υψηλών Επιδόσεων. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Ικμάντας Μπαλτσίτης. Να σας υπενθυμίσω την πρόταση της Κομισιόν για έναν ε, κανονισμό του Συμβουλίου που θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Πληροφορικής Υψηλών Επιδόσεων δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να συντάξει μία έκθεση υπό τη διαδικασία της διαβούλευσης. Πρόκειται για μία τυπική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα μπορώ να σας παρουσιάσω μια έκθεση για ένα πάρα πολύ σημαντικό κανονισμό. Η πληροφορική υψηλών επιδόσεων είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας. Ζούμε στην εποχή της γνώσης και του ανταγωνισμού και η ικανότητά μας και η γνώση μας να εκτελούμε, εξασφαλίζει τη δυνατότητά μας να εκτελούμε πολλές δράσεις σε πολλούς τομείς ε, της ζωής μας. Σήμερα η Ευρώπη χάνει τον, ε, την ανταγωνιστικότητά της ε, στον τομέα αυτό, στο παρελθόν. Είμαστε μία από τις δέκα χώρες που είχαμε πληροφορική υψηλών επιδόσεων. Σήμερα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σήμερα η Ιταλία έχει την 14η θέση παγκοσμίω και είναι 12 φορές πιο αργοί οι υπολογιστές της σε σχέση με τους υπολογιστές υψηλής ταχύτητας που βρίσκονται στην Κίνα. Έτσι λοιπόν η υψηλή ταχύτητα ε, ουσιαστικά έχει κατακτηθεί από την Ιαπωνία, την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ελβετία. Και οι υπολογιστές που έχουμε εξαρτώνται από μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες. Αυτό μας θέτει σε μία μειονεκτούσα θέση. Καθυστερούμε σε αυτόν το τομέα και αυτό μας ε, έχει θέση εκτός παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι επενδύσεις μας είναι αναπαρκής Και αυτό σημαίνει ότι είναι αρνητικός ο αντίκτυπος ε, στις οικονομίες μας επιστήμη μας και η βιομηχανία μας πρέπει να δημιουργήσει δεδομένα και υποδομές που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέτει απειλές για την ασφάλεια των δεδομένων. Εμείς δίνουμε τα δεδομένα μας σε τρίτες χώρες χωρίς να υπάρχουν εγγύσεις προστασίας των δεδομένων. Με τη διαρροή των δεδομένων χάνουμε γνώση και ανταγωνιστικότητα αλλά και τεχνογνωσία. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και επιζήμια ως προς την ανταγωνιστικότητά μας ε, Πρώτη όψεω, αν δεν ξέρει κάποιο ε, πολλά, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να κατανοήσει τις ε, ε, διαδικασίε δεδομένων υψηλών ταχυτήτων. Όμως τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε όλου τους τομείς, το χάρη στα νέα φάρμακα, στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, την καινοτομία, στην τεχνολογία, στην ιατρική, στη διάγνωση και σε εξειδικευμένες θεραπείες, στις δημόσιες υπηρεσίες, ε, τα μέσα μεταφοράς, όλα αυτά εξαρτώνται από ροές δεδομένων. Θα έχουμε τώρα μια νέα εποχή ε, με νέα φάρμακα στις αγορές. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να έχουμε πιο συγκεκριμένες θεραπείες που να είναι πιο αποτελεσματικές. Σήμερα χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να αναλάβουμε πήγουσα δράση στον τομέα αυτό. Γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν να συσταθεί μια Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Πληροφορικής Υψηλών Επιδόσεων και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των τεχνολογιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι απαραίτητο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι υποδομές υψηλών ταχυτήτων χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις και κανένα από τα κράτη-μέλη δεν μπορεί να κάνει αυτές τις επενδύσεις από μόνο του. Έτσι λοιπόν αυτή η κοινή επιχείρηση είναι η κατάλληλη πλατφόρμα. Η κοινή επιχείρηση θα προβαίνει στην ε, αγορά στις προμήθειες των ε, ε, υπερυπολογιστών και επίσης θα μπορεί να δημιουργεί τέτοια συστήματα. Η κοινή επιχείρηση θα οργανώσει κοινέ δημοπρασίες για υπολογιστές που θα λειτουργούν στην ε, προέξα κλίμακα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι μέχρι το 1921-22 να πετύχουμε το τεχνολογικό επίπεδο που θα μας επιτρέψει να έχουμε ε, δραστηριότητες στην εξακλίμακα. Παραδείγματο χάρη ε, στην 18η το δευτερόλεπτο. Ποιος θα συμμετέχει σε αυτή την ε, κοινή επιχείρηση. Έχουν υπογραφεί ήδη οι διακηρύξει κοινή επιχείρηση από 14 κράτη και η Ελβετία θα συμμετέχει ως συνδεδεμένη χώρα. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και σε άλλα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη. Το θέμα τη χρηματοδότηση έχει ω εξή. Το 50% θα προέρθει από τον προπολογισμό τη Ένωση και η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα έλθει από τις συμμετέχουσες χώρες το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προέλθει από το Μηχανισμό Συνδέοντας στην Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020. Η συνεισφορά των ε, κρατών που θα συμμετέχουν θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Η κοινή επιχείρηση δεν ε, χρειάζεται νέα κονδύλια από άλλα προγράμματα το 2018, ε, στον προπολογισμό 2018-2020 έχουν προβλεφθεί αυτά τα κονδύλια στα προγράμματα που πολύ σας ανέφερα. Η χρηματοδοτική συνεισφορά των κρατών μελών δεν αναφέρεται στον κανονισμό. Η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο της κοινή επιχείρησης και θέλω να σας αναφέρω και κάποιες άλλες πτυχές. Η πρόσβαση στην υποδομή και η προστασία των δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων θα ρυθμίζεται από τους υφιστάμενους κανόνες και όλες οι χώρες θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες αυτούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, το 50% ε, θα χορηγείται στο σύνολο των ενδιαφερομένων χωρών και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και ο Μηχανισμός Συνδέοντας για την Ευρώπη θα ισχύουν ως προς τους κανόνες. Οι κανόνες των προγραμματών αυτών θα εφαρμόζονται. Το υπόλοιπο 50% θα καταναμεθεί μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Ελπίζω να μπορέσετε να με υποστηρίξετε, συνάδελφοι, στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη έτσι που συντομεύω τη διαδικασία. Είναι σχεδόν όλοι οι σκιώδεις εδώ, ευτυχώς. Ο κύριος Μπόνι έχει το λόγο για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε, την πολύ καλή προπαρασκευή. Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε την έλλειψη των δυνατοτήτων ε, σε ό,τι αφορά την, την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, αλλά σημειώνεται πρόοδος. Ε, σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα ε, για τους στόχους της στρατηγικής μας. Ε, οργανώνεται η κοινότητα HPC για να έχουμε μια ηγετική, ένα ηγετικό ρόλο να υπάρχει πρόσβαση στην χρήση αυτών των υπερυπολογιστών και να μπορέσει να προωθηθεί και η αλυσίδα διανομής σχετική. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ε, σε αυτή την ψηφιακή ε, εποχή χωρίς να έχουμε αποδοτικά ε, δίκτυα, δίκτυα υψηλής απόδοσης ε, πληροφορικής. Ε, γίνονται προσπάθειες όπως με το δίκτυο Jang που ενώνει ήδη 50 εκατομμύρια ερευνητές. αυτή η πληροφορική υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να δίνει πρόσβαση στους υπερυπολογιστές. Και υπάρχει και ευρωπαϊκή τεχνολογία, ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα. Ε, ελπίζω αυτή η πρωτοβουλία να προσελκύσει επενδύσεις έτσι ώστε να φτάσουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς, να στους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές, να υπάρξει μια κοινή σύμπραξη η οποία έχει ως στόχο να αναπτύξει ε, συστήματα υψηλής απόδοσης έως το 2022 και το 2023. Η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή που γίνεται προς την υποστήριξη της ακαδημαϊκής ε, κοινότητας για να, για να αναπτυχθεί αυτή η σύμπραξη HSPC με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας ε, για να έχουμε υψηλή απόδοση EPP αλλά και CPP για να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα ε, να έχουμε μια οικονομία που θα βασίζεται στα δεδομένα. Ε, θα ήθελα περισσότερα κράτη-μέλη, αναφερθήκατε στα 13 βέβαια, 14, ε, θα ήθελα περισσότερα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η δική μου η χώρα, η Πολωνία, να συμμετάσχουν ε, σε αυτήν την κοινή σύμπραξη και να αποτελέσει αυτό ένα τομέα προτεραιότητα για, για προγράμματα έρευνα και ανάπτυξη ε, ε, με βάση και τις εθνικές ε, δραστηριότητες. Ευχαριστώ και τώρα κύριο Στοσανόσκη για την ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή βάση περαιτέρω εργασιών, ε, διότι υποστηρίζεται τη συνέργεια σε ό,τι αφορά ε, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα να υποστηρίξω μια άλλη καλή ιδέα τη δημιουργία αυτής της ευρωπαϊκής κοινή σύμπραξης προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω αυτή η σύμπραξη να πάρει σάρκα και οστά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλες, ε, άλλους παίχτες παγκοσμίως εγώ προείδρευσα ε, της εποπτικής, ε, του Εποπτικού Συμβουλίου μιας ε, εταιρείας καινοτομίας στον τομέα πληροφορικής για πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να σχεδιάσει κανεί ένα project και να βρει χρηματοδότηση κυρίω για να δημιουργήσει έναν υπερυπολογιστή, ένα super computer. Ανησυχώ κάπω σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση. Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι όλα θα γίνουν από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης θα είναι δύσκολο να βρούμε όλα τα συστατικά. Όταν φτιάξαμε τον υπερυπολογιστή εμείς πριν από μερικά χρόνια ήταν δύσκολο να γίνει αυτό μόνο από ευρωπαϊκές πηγές. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για εξαιρετικά εξειδικευμένο εξοπλισμό. Είναι πολύ αυστηρές, πολύ ε, ε, καταναγκαστικές αν θέλετε οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις ε, υπάρχουν και κάποια ακόμα σημεία που θα ήθελα να προσθέσω σε ό,τι αφορά την έκθεση υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι προσυζήτηση το πρώτο είναι η πρόσβαση των τρίτων χωρών εγώ θα πρότεινα να είμαστε ανοιχτοί να είμαστε ευέλικτοι εδώ Ας μην περιορίσουμε τη διεθνή συνεργασία. Δείτε τι κάνει το Ισραήλ, παραδείγματο χάρη. Μια χώρα πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τεράστιες δυνατότητες στον τομέα της γνώσης. Ε, ας μην κλείνουμε τις πόρτες μας λοιπόν. Και με βάση την εμπειρία μου στην επιχείρηση όπου εργαζόμουν, ε, είναι η αυστηρά ε, πολιτική χρήση, αστική χρήση, εν ότι είπαμε ότι αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς ε, αστικούς, πολιτικούς, αλλά και για το PRS και για τις υπηρεσίες ασφαλείας, τελικά αυτά τα πράγματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, και αλλού. Δεν θα ήμουν λοιπόν τόσο αυστηρός, τόσο ε, περιοριστικός, διότι οι υπηρεσίες ασφαλείας αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Αν δηλαδή βάλουμε τόσο στενό περιορισμό θα είναι δύσκολο να τον τηρήσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ και αναμένω περαιτέρω συνεργασία. Και τώρα από τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή του εισαγωγή και τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις θέσεις του ECR και του κυρίου Τοσενόφσκι, βλέπουμε εδώ προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Η Ευρώπη δηλαδή μπορεί να κάνει ε, περισσότερα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, ο καθένας ε, στο κράτος μέλος του. Και, ε, όπως είπε και ο εισηγητής, ήμασταν επικεφαλής σε τέτοιου τύπου τεχνολογίες πριν από μια δεκαετία, ενώ τώρα ε, καθυστερούμε. όσον αφορά νέα υλικά για οικοδομές, για την άμυνα, χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη τέτοιων υλικών υπερυπολογιστές και θα τους χρειαστούμε και στο μέλλον. Ως Κοινοβούλιο δεν συμμετέχουμε στην νομοθετική διαδικασία στο θέμα αυτό. Θα μπορέσουμε όμως να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο ότι θέλουμε να προχωρήσει το θέμα αυτό, καθώς και ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε ισχυρότερη ε, συνεργασία όταν μιλάμε για υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Επίσης, ε, περιμένουμε μια νέα σειρά εγγράφων για το, ε, πρόγραμμα πλαίσιο, για το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, δεν έχουμε λάβει σαφή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το τμήμα του προγράμματος πλαισίου που έχει να κάνει με τους υπολογιστές. Νομίζω λοιπόν ότι αν συνεργαστούμε θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα που θα έχει επιπτώσεις θετικές και για τη βιομηχανία και για ε, την ιδιωτική ζωή στο μέλλον. Ε, μόλις στην αρχή έχουμε δει, αν δεν είμαστε ε, διατεθειμένοι να κάνουμε το άλμα θα υστερήσουμε και Θα είμαστε σαν τους ε, γέρους που απολαμβάνουν ακόμα τα μετάλλια που κέρδισαν στους Ολυμπιακούς στη δεκαετία του 30. Θα πρέπει να κερδίσουμε καινούργια μετάλλια στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ η Πράσινη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Άλλα μέρη του κόσμου ε, σημειώνουν πρόοδο στον θέμα της ε, υπολογιστικής ε, πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να κλείσουμε το χάσμα και αυτή η κοινή δράση θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Ωστόσο, η δημιουργία σωστής υποδομής είναι μέρος μόνο της προσπάθειας που απαιτείται. Χρειαζόμαστε και τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια υποδομή. Κινούμαστε προς μια ψηφιακή κοινωνία και ίσως σήμερα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον καθένα βήμα-βήμα να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτήν την κοινωνία. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε και το χάσμα όσον αφορά τα δύο φύλλα στο θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες ε, στους τεχνολογικούς τομείς. Ε, Θέλουμε ε, να ζούμε σε μια ειρηνική κοινωνία και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων ε, θα είναι πλεονέκτημα σε μια τέτοια κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους που έχουμε με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Θέλουμε λοιπόν αύξηση της διαφάνειας, καλύτερη διαχείριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριο Σιλικιώτη από την ΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. <clears throat> Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σικμάντα για την έκθεση που έχει καταθέσει. Ε, η ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτικής Αριστερά ε, έχει ορισμένου προβληματισμού και ανησυχίε για την πρόταση όπω ε, προτείνεται από την Κομισιό. Είναι γι' αυτό που χαιρετίζομαι τι σημαντικέ βελτιώσει που γίνονται από τον εισηγητή τη ΙΝΤΡΕ. Για μα είναι σημαντικό η όποια επένδυση γίνει από την Ένωση στον τομέα της πληροφορικής υψηλών να έχει ως στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων της κοινωνίας. Για παράδειγμα, οι υπεροπολογιστές ε, ψηλού επίπεδου θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, στηρίζοντας ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτές ε, που αποτελούν και τον πυλώνα της οικονομίας της Ένωσης ε, ιδιαίτερα στηρίξουν για σκοπούς προσωμείωσης, απεικόνησης και πρωτοτυποποίησης. Ε, τώρα θα πω και κάποιες επιφυλάξεις. Πρώτα-πρώτα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η πληροφορική υψηλών επιδόσεων για την αμυντική βιομηχανία και για στρατιωτικούς σκοπούς ή για ε, ε δράσεις που έχουν στόχο την ασφάλεια σε εισαγωγικά αλλά στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιούνται για να παραβιάζουν ανθρώπινε πολιτικέ ελευθερίε, την ιδιωτικότητα αλλά και τα προσωπικά δεδομένα. Η δεύτερη επιφύλαξη υποχωμένη είναι, σύμφωνα με την πρόταση τη Κομισιόν, η πρόσβαση στου υπεροπολογιστέ θα είναι ανάλογη προ τι χρηματοδοτικέ εισφορέ των κρατών μελών. Θεωρούμε πω η πρόνοια αυτή λειτουργεί υπέρ των μεγάλων κρατών και σε βάρο των πραγματικών αναγκών που έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Εμεί ζητούμε να διαγραφεί αυτή η πρόνοια που προτείνεται από την Κομισιό Ε, θέλουμε να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκε για τους χρήστες από όλα ε, τα κράτη-μέλη. Ε, και ε, τέλος είναι σημαντικό πως η κοινή επιχείρηση με τους υπερπολογιστές υψηλών επιδόσεων θα συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Νομίζω και οι εμπειρίες που έχουμε στον τομέα αυτό με τεχνολογίες εχμής στο τελευταίο διάστημα ε, μας ε, δημιουργά περισσότερες έγνοιες ότι πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε μια τέτοια νομοθεσία που να προστατεύονται πραγματικά τα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή και η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το μέλλον της ψηφιακής ε, κοινωνίας ε, που αναπτύσσεται παγκοσμίω. Πρέπει να τονίσουμε ότι η πληροφορική υψηλών επιδόσεων δεν ε, σημαίνει το ίδιο με υπολογιστές υψηλών επιδόσεων. Κάποια φορά φαινόταν ε, ότι περιορίζουμε την πληροφορική υψηλών επιδόσεων ε, στην ε, τεχνολογική συνιστόσα. Όμως για να έχουμε πληροφορική υψηλών επιδόσεων πρέπει να έχουμε και άτομα με υψηλές επιδόσεις, με πολλά προσόντα και πρέπει να έχουμε διαδικασίες υψηλών επιδόσεων και πρέπει να έχουμε και αλγορίθμους βελτιστοποίησης και σε αυτές τις διαδικασίες εκμάθησης και σε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις κοινέ αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος το οποίο η ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabyte να μην έχει τις ίδιες κοινέ αξίες ή καλύτερες που έχει και ε, η ευρωπαϊκή ε, κοινωνία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μία πληροφορική υψηλών επιδόσεων που να έχει μία ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό πρέπει να υπάρχει και είναι παρόν σε όλες τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας. Να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των εννέα κοινοβουλίων της ενεργειακής κοινότητας. Εννέα χώρες από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Δυτικά Βαλκάνια. Και σε λίγο θα συζητήσουμε το θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για σας. Όμως, παρ' αυτά, τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το σημείο 14 την κοινή επιχείρηση πληροφορική υψηλών επιρρώσεων. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Τόμας Κόρτας, ο οποίος είναι διευθυντής ε, της ε, επιστημονικής υποδομής και της ψηφιακής αριστείας. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΤΡΕ για τη δυνατότητα μου δίνει να απευθυνθώ ε, σε αυτήν σήμερα. Εμείς καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Μπάλτσιτης. Ε, ακούσαμε και τα σχόλια του σχεδόν συγγητών, τα σημειώσαμε, καθώς και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και που ενδιαφέρονται για αυτήν. Χαίρομαι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναγνωρίζεται τη στρατηγική σημασία αυτού του φακέλου, δηλαδή αυτή η κοινή σύμπραξη ε, για να είναι στην πρώτη γραμμή η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ψηφιακή ολοκλήρωση ε, και τη μετατροπή της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία γνώσης και πληροφορίας. Ε, νομίζω ο κ. Μπάλτσιτης τα είπε πολύ σωστά προηγουμένω, αλλά και οι συγητές. Να σας πω απλώς ότι στο Συμβούλιο προχωρούν οι συζητήσεις για τη δημιουργία της σύμπραξης. Η Βουλγαρική Προεδρία εργάζεται έτσι ώστε να υπάρχει μια γενική προσέγγιση πριν το τέλος του εξαμήνου και ελπίζουμε και εσείς να έχετε ως τότε ολοκληρώσει την γνωμοδότησή σας. Θα αναρωτιέστε γιατί τόση βιάση. Ακούστε, μένα από τα επιχειρήματα ήδη ακούστηκαν. Όχι μόνο δεν είμαστε στο top 10, χάνουμε και την επόμενη γενιά τεχνολογιών. Ε, δεν έχουμε τις κατάλληλα μηχανήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονές μας, τη βιομηχανία μας, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και το δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν αυτού τους υπερυπολογιστέ και να μπορούν να επεξεργαστούν πάνω από 700 ε, ε εφαρμογέ που εξαρτώνται από αυτού του υπολογιστέ. Πολλέ από αυτέ τι εφαρμογέ μάλιστα αναφέρθηκαν σήμερα. Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία ήδη δημιουργούν αυτού του υπερυπολογιστέ. Ε, Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στο top 10 και το 2021 είναι ο δικό του στόχο για να έχουμε τη νέα ε, γενιά υπερυπολογιστών. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε μαζικά ε, για την επόμενη, γενιά, την επόμενη τεχνολογική γενιά. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφο, θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά τα μηχανήματα, του υπερυπολογιστέ, ταυτόχρονα ε, να επενδύσουμε στη νέα γενιά ε, τεχνολογία όπου είμαστε πίσω. Και εδώ μιλάμε για την τεχνολογία excess skills. Ε, δεν έχουμε όλες τις, α, ε, όλα τα στοιχεία για να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε ε, αυτές οι τεχνολογίες ε, της εξακλίμακας να προχωρήσουν. Θα πρέπει να ξεκινήσει η δουλειά τώρα, διότι ο νέος κύκλος για αυτές τις τεχνολογίες ε, κρατάει τουλάχιστον τέσσερα ή και πέντε χρόνια. Και η σύμπραξη δεν θα επικεντρωθεί μόνο ε, στο να έχουμε κάποιες, ε, κάποια μηχανήματα εχμής, ε, όχι μόνο για αυτές τις τεχνολογίες εξακλίμακας, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και καινούργιες καινοτόμες εφαρμογές, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις δυνατότητες καινοτομίας και να οικοδομήσουμε και να αναπτύξουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις τεχνολογίες. Είμαι σε θέση να σας πω σήμερα με χαρά ότι δεν είναι μόνο 14 κράτη-μέλη τα οποία έχουν υπογράψει τη δήλωση, ε, είναι ακόμα πολλά κράτη-μέλη τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν την κοινή σύμπραξη. Η Πολωνία, η οποία πρόσφατα είπε ότι είναι διατεθειμένη να, να, υπογράψει τη δήλωση αυτή πολύ σύντομα, το ίδιο είχε για τη Σουηδία και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και άλλα καλά νέα, όχι μόνο από, μικρές, από μεσαίες και μεγάλες χώρες, αλλά και από μικρές χώρες, διότι είναι θεμελιώδη σημασία σε αυτό να δημιουργήσουμε ίσες ε, ευκαιρίες για όλους, ένα ίσο πεδίο ευκαιριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια λέξη ακόμα, Πρόεδρε. Θέλουμε να δώσουμε το χρόνο πρόσβασης που χρειάζονται όλοι ε, στα μηχανήματα αυτά, τα οποία θα μας ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτή την ε, σύμπραξη, με αυτή την προσέγγιση 50-50. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής τώρα, ο κ. Μπαλτσίτης, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Όλα τα θέματα που εξετάζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά, όμως ε, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και στη συζήτηση για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένε ιδέες, γιατί μιλάμε για το μέλλον μας. Ε, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις βιαστικά. Η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί μια βάση για την ε, νέα μας ζωή στο μέλλον. Και θυμάμαι το 2003, όταν στη Λιθουανία συζητούσαμε τα συστήματα πληροφορικής ε, και τις ε, συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Μιλούσαμε για το πώς θα καταργούσαμε τα καλώδια. Τότε ήμουν υπουργό μεταφορών και με κατηγόρησαν ότι είχα δώσει πάρα πολύ χρήματα για αυτό το σκοπό. Όμως ε, τελικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που τελικά βάλαμε αυτά τα καλώδια και έχουμε μία από τις πιο υψηλές ταχύτητες διαδικτύου στην Ευρώπη και μπορέσαμε να δούμε τα ωφέλη μόνο μετά από 10 χρόνια. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θα μπορέσει και η Κομισιόν να παρουσιάσει όλες τις κατάλληλες απαντήσεις από σκοπιά τεχνολογίας. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα σχετίζεται με το μέλλον μας. Επομένως πρέπει να αναλάβουμε ταχύτατη δράση και να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Γιατί αυτό απαιτεί καθημερινή ζωή. Σας ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή και για την ομιλία σας. Ε, λοιπόν, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 26 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, όλα την Πέμπτη. Η ψηφοφορία στην Ήτρα 19 Ιουνίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλη είναι προ επιβεβαίωση. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ε, ημερησίας διάταξης, την ανταλλαγή απόψεων με την ενεργειακή κοινότητα. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση πριν 1,5 χρόνο μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου. Είχε εκπροσωπηθεί και η Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας και εκεί συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι από εννέα κοινοβούλια από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, η οποία ασχολείται με τη βιομηχανία, τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, την έρευνα, την ενέργεια. Και φυσικά ασχολείται μέρη και με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, το ψηφιακό θεματολόγιο, ακόμη και την διαστημική πολιτική. Έχουμε λοιπόν πολλές ευθύνες και έχουμε εμπλακεί, συγγνώμη, εμπλεκόμαστε στην πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γιάννης Κόπατς είναι επίσης εδώ μαζί μας, είναι διευθυντής της ε, γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας στη Βιέννη. Και ε, πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Σλοβενία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Διευθυντή και τα μέλη των κοινοβουλίων ε, των ε, συμβαλωμένων μερών της συνεργικής κοινότητας και να σας πω ότι η συζήτηση στην Ήτρε έχει προγραμματιστεί επί τη ευκαιρία της δεύτερης συνάντησης της κοινοβουλευτικής ονομέλειας της ενεργειακής κοινότητας. Επίσης, Πρόκειται για μια διεθνή ένα διεθνή οργανισμό όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες από την Ανατολική Ευρώπη και τον Αυξήνο Πόντο. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Διευθυντή για μια εισαγωγική παρουσίαση και Μπορούμε να δούμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις τις δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η δέσμη μέτρων στην Επιτροπή μας. Ε, στη συνέχεια θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία από συζήτηση με τα μέλη και καλούμε και τους βουλευτές της ενεργειακής κοινότητας να συμμετέχουν στη συζήτηση. Ίσως Ε, στην αρχή της συζήτηση, επειδή δεν έχετε τις κάρτες μαζί σας, ενώ εμείς έχουμε τις δικές μας κάρτες, ίσως να μπορούσατε να ε, συστηθείτε, να πείτε το όνομά σας και από ποια χώρα προέρχεστε, τίποτα άλλο. Έτσι να ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε. Να ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της ομάδας. Θα συμπροεδρεύσουμε και οι δύο. Συμπροεδρεύαμε Λέγομαι Γκουραν Μιλένσκι, ε, μέρος ε, του Κοινοβουλίου της Μακεδονίας. Λέγομαι Χάρη Λόκβενετς, μέλος ε, του Κοινοβουλίου της Μακεδονίας, παραμονός συνάδελφος, ευχαριστώ. Με μέλη Αϊτσίρη και εγώ μέλος του, του Μακεδονικού Κοινοβουλίου. Thank you. Member. Μέλος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας.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 από το Κωσυφοπαίδιο, μέλος του Συμβουλίου του Κωσυφοπαιδίου. Dardan Sidiou, member of the Parliament of Kosovo. Από το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπαιδίου. Snežana Petrović, Serbian Parliament. Από τη Σερβία. Member of the Serbian Parliament. Από τη Σερβία. Andri Hasa, member of Parliament of Μέλος του Κοινοβουλίου της Αλβανίας. Edward Chalsi, from Albanian Parliament από το Αλβανικό Κοινοβούλιο. από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Fine. Thank you for your presentation. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο λοιπόν τώρα στον κύριο Διευθυντή για να ακούσουμε την παρουσίασή του. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπούζεκ, σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε, που μας δώσατε τη δυνατότητα να ε, εμφανιστούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι ε, που δίνει νέα ζωή στην ε, κοινοβουλευτική μας συνέλευση. Ευχαριστώ και όλους τους ευρωβουλευτές που έδειξαν ενδιαφέρον να συνομιλήσουν μαζί μας και που μας αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους. Η ενεργειακή κοινότητα είναι πανευρωπαϊκός οργανισμός όπου συναντάται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις γειτονικές της χώρες. Οι γειτονικές χώρες αλλάζουν. Ε, ε, χάσαμε ε, την Βουλγαρία και την Κροατία διότι προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως έχουμε τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Η ενεργειακή κοινότητα πέρα από το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο μόνος πραγματικά πανευρωπαϊκός οργανισμός ε, όπου συμμετέχει το σύνολο της Υπήρου. Ε, οι συμβαλόμενοι, οι γαλάζιες χώρες, δεσμεύονται μονομερώς και ε, εθελουσίως να εφαρμόσουν το ενεργειακό κεκτημένο καθώς και θέματα περιβαλλοντικά και θέματα που αφορούν το κλίμα μία επισκόπηση της κατάστασης. Βλέπετε εδώ τις χώρες που ε, έχουν εφαρμόσει εν μέρη ή πλήρως ε, την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Τρεις μόλις λοιπόν από, τις, ε, από τα εννέα συμβαλωμένα μέρη δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα ε, την τρίτη δέσμη μέτρων. Η Γεωργία όχι, διότι ε, προσχώρησε ε, στον οργανισμό μας πολύ πρόσφατα, δεν είχαν το χρόνο. Η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το κάνει αυτή τη στιγμή, ενώ η Βοσνία και Ζεγοβίνη έχει κολλήσει στη διαδικασία αυτή και φέτος είναι έτος εκλογών για αυτούς, οπότε δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλές εξελίξεις όσον αφορά την αγορά αερίου και ηλεκτρισμού. Ε, οι χώρες ε, αυτές ε, συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Κατά τα άλλα, Βλέπετε στο χάρτη την περιοχή, τις χώρες που εφαρμόζουν το κεκτημένο. Και ε, θα παραθέσω τα λόγια του Ναπολέοντα που έλεγε ότι όπου ισχύει ο αστικός κώδικας ε, είναι Ευρώπη. Εγώ λοιπόν θα πω ότι όπου έχει εφαρμοστεί ε, η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια είναι Ευρώπη. Δεν φαίνεται καθαρά το κείμενο στη διαφάνεια αυτή, ούτε θα το διαβάσω αλλά ακολουθούμε την ίδια βιώσιμη πολιτική για την ενέργεια που εφαρμόζει και η Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν τους στόχους του 2020. Ε, είναι λίγο λιγότεροι φιλόδοξοι οι στόχοι μας. Ε, επίσης το ίδιο ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση για το κλίμα μόνο δεν έχουμε τους ίδιου στόχου, και αυτό έχει αρχίσει να αποτελεί πρόβλημα. Ελπίζουμε αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε φέτος, ε, συζητώντα και σχεδιάζοντα του στόχου για το 2030. Διότι συμμετέχοντας στην εσωτερική αγορά ενέργειας με δύο διαφορετικές πολιτικές όμως και με δύο διαφορετικά νομικά καθεστώτα, αυτό ε, θα θα είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και γι' αυτό θα συζητήσουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης φέτος και ελπίζουμε να τους θέσουμε σε ακριβώς τα ίδια επίπεδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσουμε επίσης τους στόχους όσον αφορά τις βιώσιμες πηγές ενέργειας ε, όπου έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ίδιο λόγο θα ζητήσουμε και τους στόχους που αφορούν το κλίμα. Δεν θα σας ε, δείξω το διάγραμμα στην διαφάνεια διότι δεν ε, έχουν αναπτυχθεί ακόμα αυτοί οι στόχοι. Το επόμενο θέμα που ήθελα να αναφέρω είναι οι εκπομπές μεγάλων μονάδων καύσης. Η σχετική οδηγία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου φέτος και όλα τα συμβελόμενα μέρη μας υιοθέτησαν εθνικά σχέδια εκπομπών. Για παράδειγμα, η Σερβία δήλωσε ότι θα κλείσει 8 ε, ε, μονάδες σε λιγνίτη μέχρι το 2024. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο στόχο για μια χώρα σαν τη Σερβία και βέβαια τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει μετά την κατάργηση του άνθρακα. Στην σημερινή Ολομέλεια είχαμε αφιερώσει τη συζήτηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον στόχο να χρησιμοποιούνται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ενεργειακή κοινότητα. Και θα ήθελα να σας περιγράψω κάποιες από τις ε, ε, κάποια από τα σημαντικά διλήμματα που αντιμετωπίζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι, σε τι διαφέρουν λοιπόν ε, οι δικές μας χώρες από τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να το υπολογίσουμε αυτό σε ακριβείς αριθμούς. Εάν χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες επιδοτήσεις ε, για τα ορυκτά κάψιμα σε σχέση με τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ήταν πολύ πιο αισιόδοξη η εικόνα. Επίσης, υπάρχει υψηλό κίνδυνος στι χώρες αυτές όσον αφορά τι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε την σύγκριση της γερμανικής ομάδας προβληματισμού Αγκόρα όσον αφορά τις διαφορές σε, ε, στο κόστος κεφαλαίου ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Η Ελλάδα είχε κόστος 11% σε σχέση με τη Γερμανία 3%. Η Γερμανία, ε, στη Γερμανία είναι πολύ πιο ε, φτηνές οι επενδύσεις από ό,τι στην Ελλάδα. Φανταστείτε στις δικές μας χώρες είναι ακόμα ε, υψηλότερος ο κεφαλαϊκός κίνδυνος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πανευρωπαϊκό ε, χρηματοοικονομικό μέσο που να μειώσει τους κινδύνους αναχώρα. Αλλιώς δεν πρόκειται να έχουμε ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η πολύ υψηλή δασμή η δασμη feed feed-in. Ε, αυτό ήταν θέμα που συζητήθηκε πολύ πριν ε, κάποια χρόνια και όλοι είχαν την αίσθηση συμπεριλαμβανομένων ε, ημών ε, ότι αυτό θα έλυνε το θέμα. Τώρα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα. Ε, έχει ασχοληθεί με το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Οι επενδύσεις ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τώρα λιγότερο δαπανηρές. Το επίπεδο ενισχύσεων όμως συνεχίζει να είναι υπερβολικά υψηλό και αυτό εμποδίζει ε, την ε, περαιτέρω χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, άλλο θέμα είναι η υποτίμηση των κρατικών ενισχύσεων. Ένα παράδειγμα από μία από τις χώρες μας. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις ε, δικές μας ε, χώρες. Ε, δεν έχει η γραμματεία μας εντολή να επέμβει με τον ίδιο τρόπο που επεμβαίνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και γι' αυτό οι κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούνται πολύ και δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς ε, από τις, ε, αρχές, ε, τις κρατικές αρχές ανταγωνισμού. Επίσης, δεν υπάρχει πολιτική μετατροπή στις θέσεις εργασίας. Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα όραμα, χρειάζεται να έχουν μια εικόνα του πώς μπορεί να αναδιαμορφωθεί το μέλλον τους. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα προγράμματα, τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα, για το πώς μπορούν οι ανθρακορίχοι να γίνουν δασοκόμοι και πώς μπορεί η βιομάζα να χρησιμοποιείται αντί για τον ε, άνθρακα ε, για να παρέχει τον βασικό όγκο ηλεκτρικής ενέργειας ε, που χρειάζεται αλλά αυτά τα επιμέρους προγράμματα χάνονται στο γενικότερο πολιτικό τοπίο. Και τέλος υπάρχει η ε, αντίσταση στην εισαγωγή ε, ηλεκτρικής περιφερειακής αγοράς. Μπορώ να σας ε, παρουσιάσω τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύσαμε πριν περίπου ένα χρόνο που δείχνει ότι στην νότιο-ανατολική Ευρώπη 271 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων θα προκύψουν ε, από το διασυνοριακό εμπόριο. Πολλοί κατεστημένοι φορείς όμως ε, στις ε, χώρες μας θέλουν να συνεχίσουν την απομόνωση των χωρών τους, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ένα μονοπόλιο. Το να έχει κανείς τη δική του αυλή. Οι κρατικές ενισχύσεις φαίνονται πολύ καθαρά σε τούτη τη διαφάνεια. Το διάγραμμα αυτό δείχνει τις τιμές ε, ηλεκτρισμού το 2017 στις χώρες μας. Και η ευθεία που βλέπετε είναι 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή είναι η τιμή στην πιο πρόσφατη ε, λιγνητική ομάδα στο Κωσυφοπέδιο, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην τιμή της αγοράς και την τιμή που υποσχέθηκαν στον φορέα εκμετάλλευση ε, με τις κρατικές εγγύησεις. Ε, κάποιος το πρέπει να πληρώσει τη διαφορά, δηλαδή οι φορολογούμενοι. Και αυτό ακριβώς δείχνει το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων πρόβλημα που είναι πολύ πιο διαδεδομένο και πολύ πιο οξύ στις ε, χώρες μας από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, θα αναφερθώ στις περιφερειακές πρωτοβουλίες. Ε, θα περάσω στην τελευταία διαφάνεια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Κάποιες από τις προκλήσεις τις ανέφερα ήδη, κάποιες όμως θα ήθελα να τις αναφέρω και τώρα. Υπάρχει έλλειψη προόδου όσον αφορά την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο σε θέματα ενεργειακά. Και αυτό αποτελεί σημείο συμφόρησης για όλη την περιφέρεια. Ε, μπλοκάρει πολλές θετικές ε, εξελίξεις διασυνοριακές στα, Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια και χρειάζεται πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές ε, για να επιληθεί το ζήτημα. Επίσης, η διαδικασία επίλυση διαφορών τη ενεργειακή κοινότητα ε, είναι επιτυχής σε μη επίμαχες περιπτώσεις. Αλλά δεν αποτελεί επαρκώς αποτρεπτικό μηχανισμό όταν διακυβεύονται πολιτικά ή εμπορικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την ε, μεταρρύθμιση της ε, σύμβασης της ενεργειακής κοινότητας. Στο, Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητάνε τα θέματα αυτά. Επίσης, οι συνάδελφοί μα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται δικά πάνω στο θέμα αυτό. Ξέχασα να τους χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ. Και θα πρέπει η ενεργειακή να λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Αρχικά αυτό ήταν ένας από τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης που παρουσιάστηκε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα πολύ σύντομα. Πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για περαιτέρω ε, ανάπτυξη της πολιτικής είναι να διασφαλίσουμε η ενεργειακή κοινότητα να μην καθυστερήσει ε, στην ε, μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Ο πρόεδρος Μπούζεκ και κάποιοι συναδελφοί σας πρότειναν οι δέσμοι μέτρων για την καθαρή ενέργεια να εφαρμοστεί και στις δικές μας χώρες έξι μήνες μετά την υιοθέτησή της. Αυτό κάποιοι το επέκριναν, κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Κάποιε εθνικέ αντιπροσωπείε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήταν κατά αυτού. Νομίζω όμω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ενεργειακή κοινότητα να διατηρήσει την ίδια δυναμική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι πολύ εύκολο να ε, διευρυνθεί το χάσμα ανάμεσα στους δύο αυτούς φορείς και δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Και τέλος, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τους στόχους του 2030. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τη διαδικασία αυτή. Αυτό όμως είναι κυρίως δικό μας καθήκον και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις εργασίες στο Υπουργικό Συμβούλιο φέτος τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ε, τις ε, ιδέες μας και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Εγώ σας ευχαριστώ έχουμε και τι προσώπους των άλλων κοινοβουλίων εδώ. Εγώ προσωπώ τον κύριο Μπούζεκ εδώ, είμαι αντιπρόεδρος, ο κύριου Χέγκελ. Είχε ένα, μια υποχρέωση ο κύριος Μπούζεκ, την οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να αλλάξει. Ε, να ξεκινήσει η συζήτηση. Τώρα έχω τέσσερις ομιλητές στον κατάλογο. Πρώτα ο κύριος Χάρη Λόκβενετς, μέλος της επιτροπή. Επιτροπής ε, ε, του Ευρωπαϊκού ΕΦΙΕΣ e από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παρακαλώ. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη του των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Νεριακής κοινότητας. Ως βουλευτής από το Μακεδονικό Κοινοβούλιο θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω κάποια πράγματα για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην δημοκρατία της Μακεδονίας. Παρά την ύπαρξη ε, θετικών συνθήκων για τη χρήση ηλιακής ενέργειας, έχουμε 250 μέρες ήλιο κατά μέσο όρο. Ε, στη Δημοκρατία της Μακεδονίας ο ήλιος δεν χρησιμοποιείται επαρκώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μερικώς λόγω της ε, πολύ ακριβής αρχικής επένδυσης για τις σχετικές εγκαταστάσεις. Ε, επίσης ε, δεν υπάρχει επαρκής ε, χρήση των λιπασμάτων. το ίδιο ισχύει και την, για τα βιοκάψιμα, το ίδιο ισχύει και για την αιωλική ενέργεια. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον, υπάρχουν μια σειρά από project που προβλέπονται. η, φάση, η δεύτερη φάση είναι το 2019-2021 και μιλάμε για ένα αεολικό πάρκο της τάξης των 15 ΜΒ για τη δημιουργία ενός νέου ε, αεολικού πάρκου 14 ε, ΜΒ αρχικά για την περίοδο 2019-2021. Οι συνολικές δυνατότητες του project θα φτάσει στα 50 ΜΒ δημιουργία ηλεκτρο, ε, ε, ε, μονάδων, χρήση της, της, των σε, είδο, σε από τον ποταμό που έχουμε εκεί. Επίσης μηχανισμοί για την δημιουργία μονάδων φωτοβολταϊκών που μπορούν να οδηγήσουν ως και 70 ΜΒ παραγωγή ε, έως το 2021. το 2020 έχουμε κάποια, κάποιες τιμές αναφοράς ε, για την αγορά ε, ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από μικρά, μικρές υδροελεκτρικές μονάδες, ε, αιωλικές, βιομάζας, βιοκαυσίμων, με στόχο να προωθήσουμε την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για να αυξηθεί η χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ενεργειακή κοινότητα και στα συμβαλόμενα μέρη μια σειρά από κίνητρα χρειάζονται έτσι ώστε να αυξηθεί η χρήση. Η χρήση πρέπει να ενθαρρυνθεί μέσω διαφόρων ενισχύσεων και ταμείων και βεβαίως θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των βιομηχάνων αλλά και των πολιτών για τις θετικές επιπτώσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι οι συναντήσεις ε, της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για διάφορα ζητήματα του ενεργειακού τομέα. Θετικά μέτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, που έχουν μάλλον, που έχουν μάλλον ε, εφαρμοστεί σε άλλα κράτη-μέλη ε, θα μπορούσαμε αυτά να τα μετατρέψουμε σε δική μας νομοθεσία και να χρησιμοποιήσουμε την επαφή μας ε, με τις επιχειρήσεις και με τους πολίτες να, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους σε ό,τι αφορά την ανάγκη μεγαλύτερης ε, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ακούω που έρχεστε από μια τόσο ηλιόλουστη χώρα. Εμείς στις Βρυξέλλες Είμαστε στην αντίθετη κατάσταση. Φαίνεται ότι πάντοτε βρέχει. Ο κύριος Ζάρκο Μίτσι, μέλος της Επιτροπής Τουρισμού, Εμπορίου και Ενέργειας από το Κοινοβούλιο της Σερβίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήτημα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, δεδομένου ότι η Δημοκρατία τη Σερβία βρίσκεται στη διαδικασία προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει πολύ μεγάλη σημασία στη, χρήση των πηγών ε, ενέργεια από ανανεώσιμε πηγές, θέλουμε να αυξήσουμε την χρήση των πηγών αυτών προκειμένου να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μέλος ε, της πολιτικής ε, που δίνουν κίνητρα, ε, όπου βασίζεται και η Σερβία όταν ορίζει τους εθνικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη το εγχώριο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μία αξιολόγηση της διάρκειας των πηγών ενέργειας από τα καύσιμα μπορούμε να αξιολογήσουμε ε, την ενέργεια από ενώσιμες πηγές. Δημιουργούνται ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα της ε, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ των ε, μελών της ενεργειακής κοινότητας. Ε, η σημαντική συνεισφορά της ενεργειακής κοινότητας μπορεί να αντικατοπτριστεί και στην ενθάρρυνση των μελών να χρησιμοποιήσουν ε, τους κοινούς μηχανισμούς συνεργασίας και την υδροδυναμική που προβλέπει η οδηγία. Επίσης, ενθαρρύνοντας την ε, χρήση ε, των αγορών ε, όπου θα καταγράφεται η προέλευση μπορούμε να συνεισφέρουμε στη μεγαλύτερη χρήση των νέων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Εντουαρτ Σαϊζή, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Εμπορικών Δραστηριοτήτων από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω αν που μας ε, καλέσατε να συμμετέχουμε στη συνεδρίαση αυτής της αξιότιμης επιτροπής και που μας δίνετε και την ευκαιρία να μιλήσουμε. Η Αλβανία έχει λαβέ πριν λίγες ημέρες μια ισχυρή σύσταση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αναγνωρίζονται οι τεράστιες προσπάθειες ε, και οι τεράστιες μεταρρυθμίσεις ε, που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά αποτελεί και μία ενθάρρυνση να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν ε, μπορούμε μία τέτοια σύσταση να την λάβουμε αν δεν έχουμε μεταρρυθμίσει την οικονομία. Και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο ενεργειακό τομέα. Έτσι λοιπόν, από μια πληπιστική κατάσταση πριν κάποια χρόνια μετακινούμαστε σε μια καλή κατάσταση όπως είναι η σημερινή. Όμως, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα αν δεν είχαμε συνεργαστεί με τις όμορες χώρες αλλά και με τους επικεφαλής της ενεργειακής κοινότητας ε, στη Βιέννη. Έχουμε ε, κάποιες αδυναμίες που μέσω του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων, της συνεργασίας, ε, της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης. Φτάσαμε σε ένα σημείο που είμαστε περήφανοι με όσο κάναμε. Και ένα δίδαγμα σε ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ, εμεί χρησιμοποιούμε πλήρω ανανεώσιμε πηγέ γιατί έχουμε ηλεκτρικές μονάδε παραγωγής που βασίζονται στο υδρόμο όντα μέλη της ενεργειακής κοινότητας. Έχουμε καλή νομοθεσία, αλλά έχουμε οικοδομήσει και ισχυρούς θεσμούς. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα αποφασισμένοι να συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι αποτελούμε συμβαλόμενο μέρος της ενεργειακής κοινότητας που είναι ένας πολύ χρήσιμος ένα πολύ χρήσιμο θεσμικό όργανο. Και πάλι σας ευχαριστούμε που μας καλέσετε να συμμετέχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λευτιλισέτσκι από την Επιτροπή Καυσίμων ε, Ατομικής Πολιτικής και Πυρηνικής Ασφάλειας από την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς ως βουλευτής ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Όσον αφορά το σύστημα μεταφοράς αερίου στην Ευρώπη. Ήταν τιμή και ευχαρίστηση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας εδώ και αρκετά χρόνια, ώστε να διασφαλίσουμε την παροχή αερίου. Και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και στο μέλλον. Ε, ενώ ο γείτονάς μας προς τα βόρειο ε, ανατολικά ε, χρησιμοποιεί το αέριο για πολιτικούς λόγους. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην αγορά ηλεκτρισμού. Γνωρίζετε ότι η Ουκρανία, το σύστημα ε, ενέργειας της Ουκρανίας συνδέεται κυρίως με την Ρωσία, ε, με εξαίρεση ένα νησί. Η αγορά της Ουκρανίας λοιπόν είναι κλειστή και γι' αυτό οι τιμές ηλεκτρισμού στο εσωτερικό της χώρας είναι από τις υψηλότερες στην ευρύτερη περιφέρεια. Και γι' αυτό θα θέλαμε να μας βοηθήσετε ώστε να έχουμε συνεργασία κάτι που θα ωφελήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την Ουκρανία. Έχουμε περίσσιο δυναμικό στην Ουκρανία. Μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ε, την ευρωπαϊκή αγορά με άλλες μορφές ενέργειας, ε, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει εμάς ε, να έχουμε καλύτερο ανταγωνισμό και έτσι καλύτερη διαμόρφωση τιμών. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι πέρσι υιοθετήσαμε νομοθεσία για την αγορά ηλεκτρισμού. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τους κανόνες αυτούς, ενώ παράλληλα ασχολούμαστε με την επικυροποίηση του συστήματος ενισχύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σκοπεύουμε να εκπληρώσουμε όλε μα τι υποχρεώσει όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στο εγγύ μέλλον. Σα ευχαριστώ για τη συνεργασία σα και σα ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθουμε εδώ. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πετζεύσκη για την παρέμβασή σα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντανταζέτσιου, πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, για τις ε, υποδομές, ε, το εμπόριο και τη βιομηχανία από το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας ε, δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εκ μέρους ε, των ε, βουλευτών που ήρθαν εδώ μαζί μου σήμερα. Το κοσυφοπαίδιο είχε αρκετά ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την ε, εφαρμογή των κανόνων και των κανονισμών που έχουν να κάνουν με τον τομέα της ενέργειας. Όπως σωστά είπε ο κύριος Κόπατς, όμως ε, έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο όσον αφορά τις σχέσεις μας με τη Σερβία. για να διασφαλίσουμε την καλύτερη ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς. Το 2016 ε, ολοκληρώσαμε τον αγωγό με την Αλβανία, που όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το 2016. Ε, παρότι ε, χρηματοδοτήθηκε από την Γερμανία. Η χρήση του αγωγού αυτού θα ωφελήσει όλη την περιφέρεια. Η Αλβανία είναι κατά 100% ε, βιώσιμη, χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, ενώ εμείς εξαρτώμαστε από το λιγνίτη θα μπορούσαμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το Λιγνίτι και να χρησιμοποιήσουμε την υδροελεκτρική ενέργεια από την Αλβανία. Στην πρωτεύουσα του Κωσυφοπεδίου έχουμε εφαρμόσει σχέδιο ώστε 90.000 πολίτες χρησιμοποιούν ατμό για τη θέρμανσή τους. Ε, επεκτείνουμε τώρα αυτό το πρόγραμμα και ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον ε, αριθμό των ανθρώπων ε, που αντί για άλλες μορφές θέρμανσης από άνθρακα για παράδειγμα να χρησιμοποιούν τον ατμό από τα λιγνητικά εργοστάσια μας, δηλαδή να έχουμε συμπαραγωγή ενέργειας και θέρμανσης. Επίσης, στο Κωσυφοπαίδιο έχουμε δώσει κάποιες πρώτες άδειες σε ιδιωτικούς φορείς για επενδύσεις σε αιωλική και φωτοβολταϊκή ενέργεια. Και ελπίζουμε ότι μέχρι το 2023 θα μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον 25 ΜΒ από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Για να έχουμε όμως σταθερό και ισορροπημένο τομέα ενέργειας είναι απαραίτητο να επιληθεί το θέμα του αγωγού που μας συνδέει με την Αλβανία. Έτσι θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη αγορά στο σύνολο της περιφέρειας και θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από την ε, συνεργασία και την ε, αλληλεξάρτηση στο σύνολο αυτής της ενεργειακής αγοράς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία να έρθουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που παρουσίασε σήμερα ο κύριος Κόπατς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, επειδή βρίσκονται εδώ οι βουλευτές από τη Σερβία και το Ξυφοπαίδιο, ίσως αυτό να συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσης μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελαν το λόγο, να κάνουν κάποια σχόλια. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Α, η κυρία Φανμπρέμπτ. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση βάσει της παρουσίασής σας που θεώρησα ενδιαφέρουσα. Πάντοτε με ενοχλεί η έλλειψη ακριβού κεφαλαίου να αποτελεί ε, λόγο να χρησιμοποιούμε αναμεινώσιμε πηγέ όπω θα έπρεπε. Εσεί αναφέρατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η κατάσταση, αν είμαστε πραγματική ένωση. Αυτή η ένωση θα έπρεπε να δρά ένα και θα πρέπει να διασφαλίζαμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη είναι προσβάσιμο το κεφάλαιο προκειμένου να δημιουργήσουμε ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Επίσης αναφέρεται τις κρατικές ενισχύσεις και νομίζω υπάρχει μία σύνδεση. Είναι σημαντικό να το ελέγχουμε αυτό το θέμα και να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδεξοι στο να θέσουμε τέλος στις κρατικές ενισχύσεις ε, ε, για το ρηκτά καύσιμα. Αυτή είναι ίσως μια ιδέα που θα μπορούσαμε εμείς ε, οι βουλευτές να την έχουμε κατά νου και να την αναφέρουμε όταν θα συζητήσουμε με την Επιτροπή, με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς και άλλους. Ίσως ε, θα πρέπει να στραφούμε σε εσά για να ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πραγματικός έλεγχος στις κρατικές ενισχύσεις με διαφάνεια και ότι θα υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στο κεφάλαιο. Γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να κάνουμε εμεί ω στιγμή αλληλεγγύη με τι όμερε χώρε. Γιατί όλοι υποφελούμαστε από μια πιο διευρυμένη ενεργειακή κοινότητα και στο θέμα της διασύνδεσης αλλά και ως προς, ε, και ως προς την εφαρμογή των κλιματικών συμφωνιών. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που θα μπορούσαμε να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Μεγκάν Ρίτσερτς, που είναι από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Σας ευχαριστώ για το λόγο. Είναι, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία να συναντηθούν τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας με τα μέλη της Ήτρε. Ακριβώς γιατί τώρα υλοποιείται τους τριμερείς διαλόγους για τρεις νομοθετικές πράξεις, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές και διακυβέρνηση στα πλαίσια της δεσμής μέτρων ε, για την καθαρή ενέργεια. Και καλούσαμε ε, πολλά από τα συμβαλόμενα μέρη για τις δραστηριότητές τους ε, ως προς τις ανανεώσιμες πηγές. Όμως είναι σαφές, όπως είπατε, ότι οι στενοί γείτονε δεν μπορούν να κλείσουν τα σύνορά τους. Η ενέργεια πρέπει να ρέει μεταξύ των σύνορων. Πρέπει να έχουμε καλές δια... Ε, διατάξεις ως ε, προς τις ενεργειακές αγορές ε, και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κοινοτικό κεκτημένο. Και φυσικά εδώ συμπεριλαμβάνονται και πολλές πτυχές που αφορούν το κλίμα. Στο πλαίσιο λοιπόν του κανονισμού διακυβερνήσεις, ε, τα συμβαλόμενα μέρη της ενεργικής κοινότητας ήδη έχουν δημιουργήσει μια ενιαία επιτροπή για την ενέργεια και το κλίμα, έχουν συζητήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να προετοιμάσουν τα δικά τους ε, εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Πρόκειται για ένα προπαρασκευαστικό έργο που προχωρά και νομίζω ότι θα πρέπει να τους τον αναγνωρίσουμε αυτό και φυσικά η γραμματεία ε, τους υποστηρίζει και επίσης αυτή ισχύει ως προς την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα τους βοηθήσει να ε, θέσουν τους δικούς τους στόχους ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ε, και την ενεργειακή αποδυτικότητα. Ήδη γίνεται πολύ προπαρασκευαστική δουλειά και θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Ήθελα να αναφέρω και μια-δυο άλλε πτυχέ που ενδιαφέρουν την ενεργειακή κοινότητα. Δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα και ξέρω ότι ο κύριο Μπούζεκ ενδιαφέρεται πολύ. Η ένα σε ό,τι αφορά ε, τι ε, περιοχέ όπου χρησιμοποιείται άνθρακα και την μετάβαση. Ε, αυτές ε, οι περιοχές θα εγκαταλείψουν την εξορρεκτική διαδικασία και το λιγνίτι. Πρέπει να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτή την βιομηχανία, από αυτόν τον κλάδο. Και επίση ε, υπάρχει και το θέμα τη ενεργειακή ανέχεια, είναι μη νομοθετικό ζήτημα και φυσικά ενδιαφέρει την ενεργειακή κοινότητα. Και όπω είπα στην αρχή, πρέπει να δούμε τη σημασία της διεύρυνσης των αγορών που συνδέεται με τις ε, γραμμές διασύνδεσης. Μια τελευταία πτυχή ως ε, προς το κλίμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο μηχανισμός παρακολούθησης και ο σχετικός κανονισμός είναι κάτι κανονικά θα έπρεπε να έχει ε, ουσιαστικά ενταχθεί στο κεκτημένο της ενεργειακής κοινότητας. Αυτό είναι κάτι που θα εισαχθεί με τον κανονισμό περί διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα δείγμα απλούστευσης διοικητικής για τα συμβαλωμένα μέρη, έτσι ώστε να γίνει αυτό άπαξ. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που ήρθατε εδώ και για τη συμμετοχή σας. Σας ε, παροτρύνω να ενδιαφερθείτε ενεργά για το έργο της ενεργειακής κοινότητας και ε, ουσιαστικά να σημειώσετε πρόοδο στον εθνικό εθιστεί όλες αυτές τις που υιοθετούμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Και τώρα ο κύριος Κόπερτς ε, για να κλείσει η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος την κυρία Βανμπρέμπτ που άνοιξε το θέμα αυτό του πανευρωπαϊσμού ε, όταν μιλάμε για την ενεργειακή αγορά. Τα συμβαλόμενα μέρη είναι μέλη της ε, ε ενεργειακής αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια κοινή προσέγγιση και από δύο πλευρές των συνόρων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια δίκτυα, έχει κάποιες οδηγίες που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη ε, να αντιδρούν ουδέτερα ε, σε ό,τι αφορά συμμετέχοντες ε, από την άλλη πλευρά των συνόρων. Τους ίδιους κανόνες έχουμε και εμείς. Δηλαδή οι συμμετέχοντες στην αγορά, τη δική μας, ε, έχουν ίσες ευκαιρίες, αντιμετωπίζουν τον ίδιο τρόπο μεταξύ των χωρών των συμβαλωμένων, έτσι, Βοσνία, Σερβία. Όμως δεν έχουν επιληθεί ε, τα ζητήματα με τον ίδιο τρόπο που έχουν επιληθεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαφορετική δηλαδή αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορετική στην Ένωση την ενεργειακή. Και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν πρέπει να μείνουν έτσι τα πράγματα. Ε, υπάρχει το θέμα της ρήτρα αμοιβαιότητα που συζητείται στο Συμβούλιο που θα, θα, υποχρεώσει και τα κράτη-μέλη στα σύνορα να, σε, να σέβονται το κεκτημένα εφόσον τα συμβαλόμενα μέρη της ενεργειακή κοινότητας σέβεται τα αντίστοιχα, ε, τις διατάξεις. Η κυρία Φαμπρέμπτ αναφέρθηκε σε ένα άλλο στοιχείο που μου έδωσε, μου δίνει ένα να πω κάτι άλλο. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε το Connecting European Facility. Είναι ένας μηχανισμός οικονομικός που χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την διασύνδεση στο εσωτερικό της Ένωσης. Ορισμένε φορές έχει ακουστεί και η ιδέα αυτό να το μοιραστούμε και για κάποια project που συνδέουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, με τρίτες χώρες, με γειτονικέ χώρες που είναι στην ενεργειακή κοινότητα αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μεγάλη όμω αντίθεση στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Όλο αυτό λοιπόν το κεκτημένο το οποίο υπάρχει, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ε, Εμεί τα σεβόμαστε όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση το σέβεται, όμως κάτι λείπει. Λείπει το CEF, Αυτό ο μηχανισμό χρηματοδότηση. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει τώρα για τη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτή η ιδέα εξίσωσης ε, ε, του κεφαλαϊκού κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει, προχωράει σιγά σιγά αυτή η ιδέα, αναφέρεται στην τελευταία εκδοχή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ίσως να είναι και η ώρα και θέλω να σας ενθαρρύνω, να ενθαρρύνω αυτή τη συζήτηση, αυτό να γίνει πανευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στο σύνολο του εδάφους του κεκτημένου που σας έδειξα προηγουμένως ε, στο χάρτη. Αυτή η πανευρωπαϊκή ε, προσέγγιση, το πανευρωπαϊκό όραμα που υπάρχει στα πλαίσια της κοινότητας ε, ενέργειας χρειάζεται να μεταφραστεί και στην πράξη με συγκεκριμένες εφαρμογές. Στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου ανέφερα κάποια σημεία ε, δεν, μπορώ, να πω ότι αυτά είναι τα συμπεράσματα βέβαια. Ε, θέλω να σας ζητήσω να υποστηρίξετε έτσι ώστε τα συμβολόμενα μέρη της ενεργείας κοινότητας ε, ε, εάν δεν γίνουν μέλη της Ένωσης τουλάχιστον να είναι ισότιμοι εταίροι στα πλαίσια της εσωτερική αγοράς ενέργειας. Αυτό το πολυμερές σχήμα δημιουργήθηκε πριν από 12 χρόνια. Τότε είχαμε την ιδέα να συμμετάσχει και η Τουρκία την τελευταία εβδομάδα των διαπραγματεύσεων η Τουρκία αποφάσισε να είναι απλά μέλος παρατηρητής και όχι συμβαλωμένο μέρος. Όμως ε, άλλες χώρες αποφελήθηκαν από αυτό το μηχανισμό ε, από την ενεργειακή κοινότητα. Ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο μια μέρα να αποφεληθεί μετά το Brexit. Είναι ε, το καλύτερο δυνατό ε, σύστημα αυτό, το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα. Αποτελεί κάποιο μέρο τη ενεργειακή αγορά τη Ευρωπαϊκή χωρί να είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάνω από το κεφάλι μα που συχνά έχει κατηγορηθεί ότι επιβάλλεται στο Βρετανικό δικαστικό σύστημα. Εν πάση η ενεργειακή ε, κοινότητα είναι ε, το κατάλληλο εργαλείο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να ενωθεί. Ε, βοηθήστε μας προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς ε, θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό και βεβαίως θέλουμε να σας βοηθήσουμε για την υποστήριξή σας η Επιτροπή Ήτρα ιδιαίτερα και ο κύριος Μπούσεκ ο οποίος πραγματικά είναι ο νονός αυτής της ιστορίας μάλιστα θα μεταφέρω τις ευχαριστίες σας προς τον κύριο Μπούζεκ. Θέλω επίσης ε, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλους εσάς ε, από τις χώρες σας. Ε, ήταν εξαιρετικά ε, χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Τώρα μπαίνουμε σε άλλα θέματα στη μέση διάταξη. Βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να κάτσετε να ακούσετε τα επόμενα θέματα που θα συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, και τώρα θα περάσουμε στο θέμα των προτύπων ε, εκπομπών, πρότυπα επιδόσεων μόνο για τι εκπομπέ από τα καινούργια πνευματικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση. Υπάρχουν νέα πρότυπα για τις εκπομπές σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από το 2020 και μετά. Ε, για αυτή τη συζήτηση η Επιτροπή ΕΝΒΗ είναι η κύρια Επιτροπή. Εμείς ε, και η Επιτροπή Μεταφορών ε, δίνουμε απλώ την άποψή μα. Ο εισηγητή θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση που αποτελείται από 36 τροπολογίε. 30 λεπτά έχουμε προλέψει για τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο κύριο ε, Ντελούντε παρακαλώ ε, να έρθει εδώ, ο Γιάκοπ Ντελούντε, να μας κάνει την παρουσίαση για 5 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Την ομιλία του 2017 για την κατάσταση της Ένωσης, ο κ. Γιούνκερ είπε ότι η αυτοκινητομηχανία της Ευρώπης πρέπει, πρέπει να, επενδύσει, να επενδύσει στο ε, καθαρό αυτοκίνητο για το μέλλον. Και για διάφορους λόγους. Είπε καταρχήν η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στα καθαρά αυτοκίνητα αν θέλει να έχει τον ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και δεύτερον, η Ευρώπη πρέπει επίσης να επενδύσει στα καθαρά αυτοκίνητα για να μπορέσει να διατηρήσει μια ισχυρή θέση στην αγορά για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το πρώτο σημείο, Κάτι σα του ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να μπορέσουμε ο τομέα των μεταφορών να συνάδει, να, ε, ε, να συνάδει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Αλλά και το δεύτερο σημείο είναι σημαντικά. Η, η, η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία μένει πίσω σε αυτή τη μετάβαση προ την κινητικότητα ε, με χαμηλή ε, χρήση άνθρακα. Αυτό είναι σημαντικό και λόγω της ανταγωνιστικότητα και για λόγους καινοτομία. Σύμφωνα με μια πρόταση μελέτη, πρόσφατη μελέτη, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούν 200.000 νέες θέσεις εργασίας εφόσον μεταφέρουμε την παραγωγή προς ε, οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Θα πρέπει εδώ να δείξουμε ηγετικό ρόλο, να, παίξουμε, να μπούμε στην πρώτη γραμμή της αλλαγής αυτής. Ο στόχος είναι το 2025 να περάσει παραγωγή προς πιο περιβαλλοντικό, περιβαλλοντικό Φιλικέ επιλογέ. πιο αυστηρά πρότυπα είναι υπέρ για τον Ευρωπαϊκό καταναλωτή από οικονομική πλευρά, ενώ τα πρότυπα για το διοξείδιο του άνθρακα οδήγησαν σε αύξηση τη τάξη ε, των 183 ευρώ για την ε, αγορά οχημάτων σύμφωνα ε, με μια μελέτη δικτύπου της Κομισιόν. Επίσης υπήρξε εξοικονόμηση, 10 δεκα, δεκαπλάσια για το πετρέλαιο και για το ντίζελ. 136.000 και 98 για το ντίζελ. Ε, αυτά μπορούν να εξηγηθούν και από τη σταδιακή αργή αύξηση ε, της, α, των, των οχημάτων μηδενικής μηδενικομπομπών. Είμαστε επίσης σχέση με την Ιαπωνία, σχέση με τον Καναδά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε στόχους που να ε, αποκρίνονται στις ανάγκες τις περιβαλλοντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επίσης έχει ένα πρόβλημα σε επίπεδο αγοράς. Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν οχήματα ε, μηδενικών εκπομπών, δεν υπάρχουν υποδομές ε, φόρτωσης. Ε, και από την άλλη δεν υπάρχουν υποδομές επειδή δεν υπάρχουν αρκετά οχήματα. Μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στην αγορά, αυξηθούν οι πράσινε θέσει εργασία και να εξασφαλίσουμε ότι θα, ρόλο, θα παίξει ρόλο αυτό ο κλάδο για να πετύχουμε του στόχου τη Ένωση. Τι προτείνουν λοιπόν οι πράσινοι. Πρώτον, προτείνουμε οι, οι μέσε εκπομπέ ε, για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα να έχουν ένα στόχο μείωση τάξη του 45% στο 2025. Στη συνέχεια θα πάμε στο 75% για το 2030. Αυτή η πρόταση μπορεί να φαίνεται ριζική εκ πρώτη όψεω όμω είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτοί οι στόχοι αφορούν μόνο τα νέα οχήματα, όχι τον υπάρχοντα στόλο. Αυτοί οι στόχοι είναι όντω φιλόδοξοι, αλλά μπορούν να επιτευχθούν και είναι και πολύ σημαντικοί εάν θέλουμε να συμμορφωθούμε με τη Συμφωνία του Παρισιού και να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή θα είναι στην πρώτη γραμμή τη καινοτομία για τα οχήματα του μέλλοντο. Δεύτερο, να προσαρμόσουμε ε, λόγω τη αποτυχία τη αγορά ε, να υπάρχει ένα ποσοστό ε, οχημάτων μηδενικών εκπομπών στον στόλο ε, για να φτάσουμε στη μηδενική, μηδενικές εκπομπές στην κινητικότητα. Χρειάζεται μια βεβαιότητα στις επενδύσεις ό,τι αφορά τις υποδομές φόρτισης για να μπορέσουμε να ε, αναπτύξουμε την παραγωγή οχημάτων χαμηλής ή μηδενικής εκπομπής. Την μελέτη ρηκτή που η Κομισιόν φτάσει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση, η αύξηση του 50% στο 2030 από οικονομικής και κοινωνική πλευρά είναι επωφελές. Η Κομισιόν όμω δεν θεωρεί ότι η δημόσια υγεία που θα ωφεληθεί το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα ωφέλη τα κοινωνικά, διότι δεν λαμβάνει την υπόψη η δημόσια υγεία μάλλον στη μελέτη τη Κομισιόν. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πραγματικά τεράστια ωφέλη με αυτόν τον υψηλό στόχο. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα για ένα λαμπρό μέλλον και για το περιβάλλον αλλά και για την ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Για να, πετύχουμε όμω αυτή ε, την, ε, το, το όφελος θα χρειαζόμαστε άμεση δράση τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που σεβαστήκατε και το χρόνο. Από το ΕΛΚ τώρα ο κύριος Σαλίνη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ότι ο συγκεκριτή μα σε όλε τι μεγάλε προκλήσει που έχουμε ενωπιών μα και στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση. Θα είμαι σύντομο. Εμείς ε, βεβαίως θα πρέπει να δεκτούμε την πρόκληση ε, του να σεβαστούμε τη συμφωνία των Παρισίων. Ε, το να είμαστε συνεκτικοί με τη Συμφωνία των Παρισίων δεν πρέπει να αποτελέσει ένα είδος πρόκλησης κατά την απόψή μας, γιατί ο εισηγητής το αιτιολόγησε, αλλά λείπουν και κάποια ακόμα στοιχεία αιτιολόγησης, τόσο χάρη, στο να ορίσουμε του στόχου αντί για το 15% το 2025 ε, λέμε για 50% το 2050 και 1 και από το 30% ε, στο 75% θα σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τέτοιους στόχους και η αυτοκινητιστική βιομηχανία θα πιεστεί τόσο πολύ και θα καταστρέψει όλους τους στόχους που έχουμε προτείνει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Ίσως θα πρέπει να δούμε την, ποιες θα είναι οι συνέπειες, ε, οι μεταβατικές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί αν έχουμε αυτόν τον διάμεσο στόχο το 2025, ε, ουσιαστικά υπολογίζουμε βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί στο ε, παρελθόν ε, και θα εκπονηθούν το 2022, ενώ το στόχο το θέτουμε στο 2025. δηλαδή θα πρέπει από το 2015 μέσα σε τρία χρόνια να φτάσουμε στο 50%. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ε, τα εργοστάσια παραγωγής, η κλάδη παραγωγής είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έχουμε και όλο τον κλάδο των προμηθευτών και μέσα σε τρία χρόνια θα έπρεπε ριζικά ε, να τροποποιήσουν ε, την βιομηχανική υποδομή τους. Όλα αυτά θα πρέπει να συνοδευτούν με τεράστια ευθύνη από την πλευρά του νομοθέτη, γιατί διαφορετικά εμείς θα γελιοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει με το Παρίσι και που προτείνουμε με αυτή την έκθεση. Υπάρχουν κάποια γεγονότα που μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μία προσέγγιση που να είναι ρεαλιστική και προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα. Το 2017 έχουμε επενδύσει, έχουμε αντιστροφή στις πωλήσει. Ε, και βλέπουμε ότι αυξήθηκε ο ρυθμός των πωλήσεων ε, αυτοκινήτων με βενζίνη. Αυτό γιατί ο καταναλωτής πρέπει ο ίδιος να ε, έχει υπόψη την πραγματικότητα και τελικά αναγκάζεται να πάρει ένα αυτοκίνητο που κοστίζει λιγότερο και μολύνει περισσότερο. Έτσι λοιπόν εμείς προκειμένου να είμαι πιστοί στους στόχους του Περισσιού, ε, όμως ε, θα πρέπει στις συζητήσεις μας να είμαστε ρεαλιστές και όχι ονειροπόλοι. Σας ευχαριστώ ο κύριος Πούπα για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Οι στόχοι που προτείνονται είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι Μέχρι τώρα έχουμε μόνο 4% ε, πωλήσει σε οχήματα που έχουν χαμηλέ ή μηδενικέ εκπομπέ. Και όταν μιλήσουμε για μηδενικέ εκπομπέ, μιλάμε για πωλήσει μόνο 1%. Έχοντας λοιπόν κατά νου την υλοποίηση αυτών των στόχων της μείωσης των εκπομπών από τους παραγωγούς, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αυτό εξαρτάται από μεγάλο βαθμό <laughs> και από την αποδοχή των καταναλωτών. Ε, γιατί αυτό συνδέεται ε, με το εισόδημα ε, του κάθε καταναλωτή, αλλά φυσικά και από την κάμερα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θα πρέπει λοιπόν να επηρεαστεί ο κατανοητής και θα χρειαστούν πολλά περισσότερα από την ενημέρωση των κατανοητών. Σίγουρα θα χρειαστούν και υποδομές ε, φόρτισης αλλά και άλλα κίνητρα οικονομικά. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία προς αυτή την κατεύθυνση μέσω φορολογικών κινήτρων όπως ε, και ε, να υπάρξει και συνεργασία με τα πολυτεχνία για να ε, προωθηθούν ε, διάφορες επιστήμες όπως η ψηφιοποίηση, η μικροελεκτρονική, η πιστοποίηση των αυτοκινήτων κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και από τη σκοπιά του κόστους που θα έχει η πρώτη φάση της ανάπτυξης και της αγωγής αυτών των νέων τεχνολογιών. Είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα στους παραγωγούς για το τι θα θέσουν στην αγορά. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριε Πούπα, ο κύριο Στοσενόφσκι, παρακαλώ. Από το ECR. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο κειμένου. Είναι πολύ φιλόδοξο το κείμενό σας. Ας έχουμε κατά νου ότι η αυτοκινητοβιομηχανία ε, είναι ένας από τους βασικούς κινητήρες της ευρωπαϊκής οικονομίας. 12 εκατομμύρια ανθρώπων εργάζονται ε, απευθείας ε, στην ε, βιομηχανία αυτή. 40 δισεκατομμύρια είναι οι επενδύσεις και για τις έρευνες και εάν έχουμε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους Αυτό μπορεί να καταστρέψει το οικονομικό μοντέλο με όλες τις σχετικές συνέπειες. Η πρόταση ασχολείται αποκλειστικά με τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, αλλά στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να βρει έναν ισορροπημένο τρόπο να μειώσει όλες τις εκπομπές, να μην επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο διοξίδιο του άνθρακα, να μην ξεχνάμε τα οξύδια του αζότου. όπως συνέβη στο παρελθόν. Το Dieselgate και οι σχετικές έρευνες ε, το κατέδειξαν αυτό. Η τεχνολογική ουδετερότητα είναι επίσης ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας κάνω έκκληση. Στην πρόταση αυτή κινούμαστε προς την κατεύθυνση των ηλεκτρικών οχημάτων, ξεχνάμε όμως άλλες τεχνολογίες. τεχνολογίες που μπορεί τελικά να κερδίσουν αυτή την ανοιχτή μάχη. Η πολιτική οι διοικήσει, οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να ευνοήσουν μία τεχνολογία εις βάρος άλλων. Είναι κακό ε, αν η πολιτική είναι υπέρ μιας τεχνολογίας ε, ενώ η βιομηχανία είναι υπέρ μιας άλλης. Και ας επανέλθουμε σε κάτι που είπανε πριν λίγο οι συνάδελφοι. Είναι φιλόδοξος ο στόχος του 30%. Κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. 30% είναι πάνω από αυτά που υποδεικνύει το ε, πακέτο η δέσμη μέτρων για το κλίμα. Θα ήθελα να είμαστε ρεαλιστικοί και να λάβουμε υπόψη μας τι είναι τεχνολογικά εφικτό, να μην ακολουθούμε μόνο τις πολιτικές μας φιλοδοξίες. Του του λεχθέντος ε, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε δεσμεύσεις ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία, να μην υπερβάλλουμε όμως, ε, διότι ε, μπορεί να μας έρθει μπούμεραγκ. Σας ευχαριστώ κύριε και ο κύριος ε, Ρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συγητή για το έργο του. Δύο γενικά σχόλια θέλω να κάνω. Παρά τον τίτλο της έκθεση αυτή, θίγει τρία θέματα ταυτόχρονα, δηλαδή ένα περιβαλλοντικό ε, ζήτημα, κλιματικό και ανθρώπινη υγεία, ένα τεχνολογικό θέμα σε σχέση με τις καλύτερες τεχνολογικές ε, επιλογές για τα μελλοντικά έτη και μια οικονομική σκοπιά, πώς θα ε, μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Ευρώπη και αυτού του συγκεκριμένου κλάδου. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει κάνει αυτό η έκθεση. Η δεύτερη παρατήρηση η πολύ μεγάλη κλίση ε, προς τις ε, εκπομπές, προς τις μηδενικές εκπομπές. Ε, εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε ο παγκόσμιος συλλογισμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ούτε το γεγονός ότι ακόμη και το 2030 η ενέργεια θα προέρχεται κατά το ίμιση από μία ανανεώσιμες πηγές. Επίσης δεν αναφέρονται κάποια θέματα στην ε, έκθεση αυτή, όπως κοινωνική αξία των εκπομπών. Αν ε, ε, δείτε το κόστος των εκπομπών σε ένα επιβάτη ένα χιλιόμετρο, δεν είναι το ίδιο με το να έχετε τέσσερις επιβάτες ένα χιλιόμετρο. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, όπως ε, και η αύξηση της ε, αυτονομίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θα πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό μας σε σχέση με τις ε, υποδομές φόρτισης. Πρέπει να δούμε και πόσα χιλιόμετρα αυτονομίας θα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε απλώς να καταργήσουμε την αιρεσιμότητα. Έτσι λοιπόν, συνολικά ε, ο συντάκτης της ε, έκθεσης Ήτρε έχει πιο ριζοσπαστική θέση ακόμη και από τον ε, εισηγητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε το εξή, να έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση και μια λογική έκθεση και να λαμβάνονται υπόψη τρεις πτυχές. Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι αντικείμενο υπεράσπισης, γιατί φυσικά συνάδει με τις οικονομικές ικανότητες και με τις περιβαλλοντικές μας στόχους. Και κλείνω λέγοντας ότι σίγουρα προσπαθούμε να είμαστε κοντά ε, στους στόχους της COP21, όμως ε, η αποστεριόρη ε, ουσιαστικά επανα προσέγγιση δεν είναι απαραίτητα μία ε, επιλογή που θα είναι σόφρον. Ίσως λοιπόν ε, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο για να είναι αποδεκτό. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Για την ΚΟΕ, ο κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Γιάκοπ Νταλούντε για την γνωμοδότηση που έχει καταθέσει το σχέδιο θέτοντα ένα θετικό πλαίσιο κατά άποψή μου για ουσιαστικό διάλογο. Η ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά συμφωνεί πω είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη του γενικότερου στόχου που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προστασία του περιβάλλοντο, ώστε να τεθεί ένα φιλόδοξο πλάνο για τη μείωση των εκπομπών των καινούριων επιβατικών οχημάτων αλλά και των ελαφρών οχημάτων. Ωστόσο, οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ε, να είναι ρεαλιστική με βάση όλα τα δεδομένα ε, στη βιομηχανία αλλά και τις προοπτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, στην Ένωση και διεθνώς. Δηλαδή πολλές φορές όταν θέτουμε στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί μπορούμε να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Όσον αφορά του καταναλωτέ, θεωρούμε απαραίτητα να διασφαλίσουμε πω θα έχουν ε, ευκολολόγητε συγκρίσιμε και αξιόπιστε πληροφορίε στι επισημάνσει σχετικά με τι εκπομπέ των αυτοκινήτων και την πραγματική κατανάλωση καυσίμων. Και επίση θεωρούμε θα πρέπει να λάβουν υπόψη τι επιπτώσει που ενδέχεται να υπάρξουν στου εργαζόμενου. Είναι ζωτική σημασία να προληφθούν οι όποιε επιπτώσει μπορεί να υπάρξουν στην εργασία με στοχοθετημένα προγράμματα στήριξη και εκπαίδευση των εργαζομένων σε συνεργασία πάντοτε με του κοινωνικού εταίρους. Ε, θεωρούμε σημαντικό ότι ε, να προωθεί η εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών για την επαναφόρτιση, παραδείγματο χάρη των αυτοκινήτων, των ηλεκτρικών, και τα κράτη-μέλη να στηριχτούν από την Ένωση ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε δημόσιε επενδύσει για αυτέ τι απαραίτητε υποδομέ. Όμω εδώ πρέπει να σημειώσω, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλε τι προσφερόμενε τεχνολογικέ επιλογέ. Θεωρώ ότι πολλέ φορέ, όπω εξελίσσεται η τεχνολογία, είναι λαθασμένο και αδόκιμο ε, να δώσουμε όλο το βάρος ε, στα ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα γιατί υπάρχουν σήμερα περισσότερες επιλογές και στο μέλλον μπορεί να έχουμε ακόμα και άλλες. Τέλος, ένα βασικό στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί είναι η ανάγκη οι μετρήσει για τις εκπομπές. Πώς πρέπει να πραγματοποιείται δηλαδή η αξιολόγησή τους και αυτό πρέπει να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες δρόμου. Η ελέγχη να είναι συνεχής και ιδιαίτερα με την έγκριση ε, καινοτόμου τεχνολογίας. Έτσι θα αποφύγουμε στο μέλλον σκάνδαλα τύπου που είχαμε στην ε, εκπομπέ αερίου στην αυτοκινητοβιομηχανία ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και προ αυτήν την κατεύθυνση θα είναι και οι, τεχνο, που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Mr. And now we have... Ευχαριστούμε τον κύριο Σιλικιώτη. Και τώρα έχουμε έξι βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να σεβαστείτε το χρόνο σας για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο, κύριε Φανμπρέντ. Θα προσπαθήσω να με συντομία. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον εισηγητή, αλλά και τους σκιώδες όλοι αναφερθήκαν στη Συμφωνία των Περισσίων και ότι θα πρέπει να τη σεβαστούμε και στη συνέχεια αναφέρθηκαν διάφορα επιχειρήματα γιατί θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με την πρόταση της Κομισιόν, το χάρη. Όλοι ξέρουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι τόσο αδύναμη ω προς τι φιλοδοξίες της που δεν θα μπορέσει να σεβαστεί του στόχου τη Συμφωνία των Περισσίων και το σημαντικό για αυτή την Επιτροπή είναι όχι απλώ ε, να έχει κατά νου τη Συμφωνία των Περισσίων αλλά και τη βιομηχανία. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ε, θα ε, συμμετέχει ισότιμα κάθε τμήμα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν εδώ μιλάμε και για ένα ισότιμο μερίδιο. Είναι πολύ σημαντικό η αυτοκινητοβιομηχανία να θέσουμε, για την αυτοκινητοβιομηχανία να θέσουμε πολύ φιλόδοξους στόχους και για την ε, ε, μείωση των εκπομπών έχουμε και πολύ χαμηλές εκπομπές αλλά και μηδενικές εκπομπές αλλά και για τη σταδιακή εξάλληψη. Να προσπαθήσουμε να βρούμε την πλειοψηφία έτσι ώστε να είμαστε πιο φιλόδοξη από την πρόταση της Κομισιόν στους δύο στόχους που θέλουμε να θέσουμε, να είμαστε φιλόδοξοι και για την εντολή για τις χαμηλές εκπομπές και επίση ε, είχαμε μια εξεταστική επιτροπή σε αυτό το κοινοβούλιο που εργάστηκε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ευρία πλειοψηφία. Θυμάστε κύριε Χένκελ, είχαμε ευρία πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για την υποστήριξη της ε, έκθεσης της Επιτροπής Dieselgate και όλοι ψήφισαν ε, να εξαλειφθούν μέχρι το 2035 όλα τα αυτοκίνητα ε, που εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι θα ακολουθήσουμε τη στάση που είχαμε στην Επιτροπή της Ελληνικής και στην Ολομέλη. Ευχαριστώ επόμενη μιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και χαίρομαι που τώρα στην Επιτροπή Βιομηχανίας ξεκινάμε τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Θα συμφωνήσω με την Καθλίν Φαν Μπρέμπτ. Φυσικά πρέπει να κάνουμε πολλά για να ε, πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα που έχουμε θέσει εμείς ήδη. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και τις ε, βιώσιμες πηγές ενέργειας ε, και την ηλεκτροκινητικότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν υψηλά κατόφλια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, δυνατότητες ιδιωτικών επενδύσεων στην, στις υποδομές, διότι χρειάζονται ασφάλεια των επενδύσεων. Να γνωρίζουν δηλαδή ότι τα αυτοκίνητα αυτά θα έχουν, τα καινούργια αυτοκίνητα θα έχουν και την ε, απαραίτητη ζήτηση. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να επιλέγει κανείς αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέρος των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραγωγούς, για, σε κατασκευαστές, για να στηρίξουμε τις υποδομές. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στο ότι αυτή η μετατροπή θα έχει και ανεπιθύμητες κοινωνικές επιπτώσεις, ε, για παράδειγμα ε, την ε, μείωση θέσεων απασχόλησης στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν και με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συζητήσουμε τα θέματα αυτά όσον αφορά ε, το, την αλλαγή του κλίματος. Αυτό αποτελεί ένα έργο μαμούθ, ένα καθήκον μαμούθ για το σύνολο της ε, κοινωνίας. Ε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες μέχρι τώρα έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, όλα αυτά να γίνουν προ αυτών ε, που έχουν ασχοληθεί με το όλο πρόβλημα. Και όσον αφορά ε, τους στόχους του 2030, είναι φιλόδοξοι οι στόχοι αυτοί και θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές ε, και ε, την ε, κατασκευή νέων οχημάτων και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Σας ευχαριστώ. Προσβλέπω στην συνέχιση της καλής συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι συζητήσαμε την οδηγία που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Και λέγαμε, χρειάζονται όλες οι θέσεις πάρκινγκ στα κτίρια, ε, όλες οι συνέστησεις θέσεις πάρκινγκ να προβλέπεται με 20%, 10%, 50%. Και λέγαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα έρθει ο καιρός που θα συζητούμε για τα αυτοκίνητα και θα είναι και ηλεκτρικά και θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε δίκτυα φόρτισης για τα αυτοκίνητα. Και πέρασε απλώ ένα χρόνο και φτάσαμε ακριβώ σε αυτή την κατάσταση που είχαμε προβλέψει πέρσι. Γιατί τότε αρνηθήκαμε να βάλουμε ε, υποχρεωτικές διατάξεις και τώρα λέμε ποια θα είναι η δική μας φιλοδοξία για το 2030 κτλ. Ιδέα δεν έχουμε. Εγώ ξέρω όμω ότι εφόσον λείπουν τα δίκτυα φορτίση δεν μπορούμε να συζητούμε ούτε για 5% ηλεκτρικά αυτοκίνητα γιατί κανένα δεν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν πιστεύω καταρχήν αυτή η οδηγία θα πρέπει να συμφωνήσει με υποχρεωτικά ποσοστά για δίκτυα φόρτιση γιατί διαφορετικά συζητούμε τελείω μη ρεαλιστικά πράγματα και πρέπει να δούμε και ποια είναι η δική μας ικανότητα ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράγουμε ιδέες που να ε, μην θεωρούνται ε, στα όρια του φανταστικού ή χιουμοριστικές. Δεύτερο, θα πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε το κίνδυνο να προσδιορίσουμε εκ των προτέρων, να προκρίνουμε τη νέα τεχνολογία. Δεν υπάρχει τώρα καμία τεχνολογία που να θεωρείται όριμη ή βιώσιμη και να μιλάμε για ποσοστά που να ξεπερνούν το 10% του στόλου των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή και ακριβώς και γι' αυτό είδα και την ιδέα ε, του εισηγητή να αποκλείσει τεχνολογίες σε περίπτωση που βασίζονται στο υδρογόνο. Είναι τεράστιο λάθος. Πρέπει να υποστηρίξουμε καταρχήν όλες τις τεχνολογίες και να δούμε ποια από αυτές αποδειχτεί βιώσιμη, εφόρος σε αυτόν τον ε, ανταγωνισμό. Και τρίτο σημείο. Πιστεύω ότι σε αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να θέσουμε την ερώτηση και στην Κομισιόν ποιε είναι οι μελέτες αντικτύπου για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τις διάφορες επιλογές ε, και να δούμε ποια είναι η πιο αληθής δυνατότητα. Παραδείγματο χάρη, πόσο μπορούμε να πετύχουμε το στόχο τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, πόσο τη εκατό θα πρέπει ε, να έχουμε, ε, τι ποσοστό αυτοκινήτων ε, μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να έχουμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Εγώ δεν πιστεύω ε, 100, 100 στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ίσω ε, αυτοκίνητα, ίσω μια υβριδική λύση να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε έναν ορίζοντα και να υπάρξει και μία λύση θαύμα που θα εμφανιστεί το 2030. Πρέπει όμως να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις που θα έχει κάθε κράτος μέλος για τα δίκτυα φόρτισης. Είτε μιλάμε για υδρογόνο, είτε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είτε για άλλες λύσεις που είναι αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμών. Νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, η γερμανική αυτομηχανία ε, θέλει να δοκιμάσει την λύση ε, με το υδρογόνο. Όμως αν η λύση που θα θετήσουμε δεν θα φέρει την υποχρέωση να δημιουργηθεί αυτή η υποδομή, θα μείνουμε ε, μόνο στην ιστορία ότι μιλήσαμε πολύ για κάτι που δεν μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί τη στιγμή που έπρεπε δεν πήραμε τα απαραίτητα μέτρα. Και εγώ σα λέω ότι πρέπει το χάρη πέρσι, λυπάμαι που απορρίψαμε αυτό το στοιχείο ε, στα πλαίσια της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και λέγανε διάφοροι, α, το 50% είναι τοπικό κτλ. Τώρα, είτε μιλάμε για υδρογόνο είτε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ε, δεν ε, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει αυτή, αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ, ο κύριος Μαρτάν. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να μην φοβόμαστε την πρόοδο, να μην φοβόμαστε να επιταχύνουμε. Και σε αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Και αυτό είναι κάτι που λειτουργεί, έτσι. Η Ρενό ανακοίνωσε μόλι ότι έω το 2022, αύριο δηλαδή, θα μπορούν να προσφέρουν 8 νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το Volkswagen έω το 2030 θα μπορεί να προσφέρει όλη την γκάμα των αυτοκίνητων της, σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πολλές αυτοκινητομηχανίε είπαν ότι από το 2030-2040 όλοι οι θερμικοί, οι θερμικοί κινητήρες θα απαγορεύονται στις πόλεις. Το λένε χώρες, μέλη αυτό. Ε, λειτουργεί αυτό λοιπόν. Και συμφωνώ και με αυτό που πάνε κάποιοι συνάδελφοι. Πρέπει να επενδύσουμε με δημόσιε επενδύσει στις υποδομέ. Και εδώ η Κομισιόν θα μπορούσε να προτείνει αυτέ οι δημόσιε επενδύσει να αφαιρούνται από το δημόσιο χρέο. Διότι και αυτό θα είναι ένα κινητή, μια κινητήριο δύναμη για τις επενδύσεις. Και εκεί που συμφωνώ επίσης είναι το θέμα ε, της τεχνολογικής ε, ποικιλομορφία. Πρέπει να σπρώξουμε για καινοτομία στη βιοκαύσιμα, στην εθανόλη, στο μα στην εθανόλη, στην τρίτη γενιά, όπου θα μπορούμε να βρούμε νέα καύσιμα με μηδέν εκπομπές ε, στο μέλλον και βεβαίω τη δυνατότητα να παράγουμε το σύνολο της απαραίτητης ενέργειας. Ξέρετε, ο μέσος όρος των ε, καθημερινών μετακινήσεων είναι 25,2 χιλιόμετρα τη μέρα. 25,2 χιλιόμετρα τη μέρα. Υπάρχουν υποδομές που προτείνουν το βράδυ όταν γυρίζουμε, αντί να βάζουμε τα αυτοκίνητα να φορτίζουν, το υπόλοιπο της μπαταρίας να χρησιμοποιείται ε, για να φορτίζει κανείς το σπίτι του και μετά να φορτίζουμε τη νύχτα. Ε, επειδή λοιπόν φτάνουμε στα ωριά μας, αυτό μας οδηγεί, μας υποχρεώνει να δείξουμε επινοητικότητα και συμφωνώ με αυτό που είπε ο σχετικά. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι κάπως ανήσυχη με την γνωμοδότηση του εισηγητή για διάφορους λόγους. Βεβαίως συμφωνώ με τη φιλοδοξία και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών ε, διευσίδου του άνθρακα, όμως ε, δεν θα έχουμε αύριο μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν ζητήματα αγοράς, ζητήματα υποδομών, θέλουμε να γίνουν όλα τα πεζοδρόμια μας ε, να είναι γεμάτα σημεία φόρτισης. Το σύστημα των πόνους εδώ επικεντρώνεται υπερβολικά σχεδόν αποκλειστικά στα υβριδικά τα οποία ε, φορτίζονται. Δεν λαμβάνουν υπόψη άλλα υβριδικά ή το, το, τα οχήματα υδρογόνου. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια πιο, να έχουμε μια, μια, μια πιο ουδέτερη τεχνολογικά στάση. Δεν είναι αυτό τώρα στόχο του 2030, αλλά με ανησυχεί ο στόχο του 2025. Ε, δεν θα γνωρίζουμε ποιε είναι οι εφαρμοστέ αξίε μόνο το 2022. Τρει μέρε δηλαδή πριν, τρία χρόνια μάλλον πριν το 2025. Ενώ η κύκλη βιομηχανική χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Τέλο, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των οχημάτων. Τα οχήματα, τα ταγιοταχή, τα ε, ελαφρά οχήματα ε, μεταφορών. η πρόταση της Κομισιόν εμένα μου φαινόταν βεβαίως βελτιώσιμη, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ισχύει το ίδιο με την γνωμοδότηση του εισηγητή που κατά τη γνώμη μου είναι κάπως δογματική. Μακριά από την πραγματικότητα του κλάδου ε, την οποία όμως ε, δεν μπο, την οποία δεν μπορεί να αγνοεί σε καμία περίπτωση η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Και τώρα Ράδιο Λουξεμβούργο, ο κύριος Τούρμες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συντάσσω την επόμενη έκθεση, οπότε θα είμαι σύντομος. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες πίσω από κάποιες τεχνολογίες. Το υδρογόνο είναι τρεις φορές λιγότερο αποτελεσματικό από την ηλεκτρική ενέργεια. Για ένα όχημα υδρογόνου χρειάζεται, τριπλάσια ενέργεια. Διότι χρειάζεται ηλεκτρόληση για την παραγωγή της στην αυτοκινητοβιομηχανία, αυτοί που λένε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνθετικά καύσιμα, εκεί πολλαπλασιάζουμε επί 8 ή επί 10. Το ηλεκτρικό όχημα λοιπόν, το ηλεκτρικό αυτοκίνητα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικό από τις άλλες αναλλακτικέ. Θα προκύψουν βεβαίως οχήματα υδρογόνου. Αλλά η φυσική μας λέει ότι κυρίως θα έχουμε ηλεκτρικά οχήματα. Και Ντομινίκ, όταν λες ότι δεν είναι σαφή τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον άνθρακα και τον απολογισμό, δεν ξέρω να γνωρίζει, αλλά γίνεται μια απέντηση στη Σουηδία για μια πρώτη γενιά πράσινης, πράσινης μπαταρίας ευρωπαϊκής, 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές οι μπαταρίες θα είναι 100% ανακυκλώσιμες με κοβάλτιο, νικέλιο που θα προέρχεται από τη Σουηδία σε ορυχεία δηλαδή που θα έχουν και ένα σήμα βιωσιμότητας ε, αν προέρχονται από εκτός ένωσης δηλαδή μη φανταστείτε τις μπαταρίες όπως τις, ε, τις γνωρίζαμε στο παρελθόν μιλάμε για μπαταρίες που θα έχουν ε, άλλα ενεργειακά δεδομένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει ένα σήμα ευρωπαϊκό για τις πράσινες μπαταρίες ακριβώς επειδή σε επίπεδο βιομηχανικό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι σε σχέση με την Ασία είναι να πάμε προς τις μπαταρίες του αύριο, τις πράσινες μπαταρίες δηλαδή. Θέλουμε να το υποστηρίξουμε αυτό, να το πλαισιώσουμε με ένα label, με ένα σήμα για να προστατεύσουμε ακριβώς ε, την ε, ε, αναδιόμενη αυτή αγορά. Επίσης ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ακόμα και στον οργιακό μίξ σημερινό, τον ενεργειακό μείγμα, είναι πέντε φορές πιο αποτελεσματική από ένα αυτοκίνητο με βενζίνη ή με δίζελ. Ακόμα και με το παρόν ενεργειακό μείγμα υπάρχει πλεονέκτημα. Και για να αυξηθεί αυτό το πλεονέκτημα στην οδηγία για τα ανανεώσιμες που διαπραγματευόμαστε λέμε σαφώς ότι θα είναι η ανανεώσιμα, η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που θα φορτίζει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι σαφώς υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων ε, η οργάνωση που βάζουμε σε θέση αυτή τη στιγμή, που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή. Yes, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λόγια. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό το θέμα αυτό και ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις όταν προσπαθούμε να μειώσουμε τις εκπομπές στις μεταφορές, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο μόνος τομέας όπου αυξάνονται συνεχώς οι εκπομπές. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ε, μεγάλες προκλήσεις και ξέρουμε ότι αυτό θα απαιτήσει και πολύ χρόνο. Δεν είναι εύκολο να μειώσει κανείς γρήγορα τις εκπομπές. Ε, μόνο τέσσερα κράτη-μέλη ε, έχουν τώρα λιγότερες εκπομπές από ό,τι είχαν το 1990 και η χώρα μου η Φιλανδία είναι μία από αυτές. Στις περισσότερες χώρες όμως οι ε, εκπομπές αυξάνονται συνεχώς και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, να μην επικεντρωθούμε σε μια τεχνολογία μόνο, διότι θα απαιτήσει χρόνο μέχρι να έχουμε νέα οχήματα. Ε, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να έχουμε βιώσιμα καύσιμα ε, στα υπάρχοντα οχήματα. Ταυτόχρονα είναι πολύ θετικό ότι προωθούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και εδώ υπάρχουν εμπόδια. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η βιομηχανία ε, συσσωρευτών ε, δεν ε, είναι αρκετά ανεπτυγμένη ακόμη και υπάρχουν και νέες τεχνολογίες όπως είναι το υδρογόνο, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία προσέγγιση τεχνολογικά ουδέτερη και κατόπιν η αυτοκινητοβιομηχανία και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι ε, θα μπορέσουν να αποφασίσουν ε, ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία. Ε, ούτε θα πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στα καύσιμα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ένα από αυτά φυσικά είναι το σύνολο της υποδομής και το σύστημα εφοδιασμού, ο σχεδιασμός του συνολικού συστήματος μεταφορών υπάρχουν πολλοί τομείς και θα πρέπει να εργαστούμε σε όλους τους τομείς αυτούς διότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τεχνολογικά οδετήρη προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ρόνο Μέτσελ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα έπρεπε να εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γιατί τα νούμερα που σας δίνουμε είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που βλέπουμε στο σχέδιο ε, έκθεσης ε, του εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει τρεις πτυχές από κοινού. Τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, τον αντίκτυπο για τον καταναλωτή και τον κοινωνικό αντίκτυπο στην απασχόληση και ιδιαίτερα ε, όσον αφορά την πτυχή της καινοτομία. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, πολλοί μίλησαν για την Συμφωνία του Παρισιού και πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές της ε, μέχρι το 2030 κατά τουλάχιστον 40% σε σχέση με το 1990. Ε, και αυτό σημαίνει ότι εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές κατά 30% σε σχέση με το 2005. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα οδικών μεταφορών, που μάλλον δεν είναι και ο πιο οικονομικός τρόπος ε, να μειώσουμε τις εκπομπές, ε, ε, η 25% θα ήταν η οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα φτάσουμε το 22%. Με μία πρόταση λοιπόν μόνο δεν θα πετύχουμε το στόχο μας όσον αφορά τις εκπομπές στον τομέα των μεταφορών. Οι υπόλοιπε μειώσεις θα γίνουν με πρότυπα διοξιδίου του άνθρακα για τα φορτηγά που ε, τον Μάιο, ε, πρόταση που θα υποβάλει τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχουμε και άλλες πολιτικές που θα συμβάλλουν στην μείωση. Για παράδειγμα, την αναθεώρηση της εροβινιέτας, ε, την, στις οδηγίες για τις συνδυασμένες μεταφορές και πολύ σημαντικό είναι το θέμα που επεσήμαναν διάφοροι ευρωβουλευτές ε, που είναι ε, οι οδηγίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για, τις, για τα μείγματα καυσίμων και τα κράτη-μέλη θα έχουν δικές τους εθνικές και τοπικές πολιτικές, διότι όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας δεν νομίζω ότι οι Βρυξέλλες είναι ο κατάλληλος φορέας. Όσον αφορά λοιπόν τις δυνατότητες για ε, υψηλότερες μειώσεις, το 40%, όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό θα σημάνει μείωση ε, τριών ποσοστιαίων μονάδων. Δηλαδή, αν ανέβουμε πιο πάνω, πάλι δεν θα έχουμε σημαντική συμβολή. Όσον αφορά ε, την εξοικονόμηση για τους καταναλωτές, ο στόχος του 30% το 2030 ε, θα σημάνει ε, εξοικονόμηση 1.400 ευρώ για τους καταναλωτές. Εάν αυξήσουμε το στόχο αυτό όμως, το όφελος για τον καταναλωτή θα μειωθεί βαθμιαία. Με αύξηση λέει, του στόχου στο 40% μειώνεται κατά 400 ευρώ, ενώ αν έχουμε το στόχο του 50% έχουμε μείωση κατά 1.000 ευρώ. Διότι το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί όσον αφορά τον αντίκτυπο στην απασχόληση. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που συζητιέται. Και έχουμε δει πολλά διαφορετικά στοιχεία πάνω στο θέμα αυτό από πολλές διαφορετικές μελέτες και θα πρέπει κανείς να εξετάσει πολύ προσεκτικά ε, τις προϋποθέσεις των μελετών αυτών στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το 30% δεν θα υπάρξει μείωση ε, στην απασχόληση. Αντιθέτω, μπορεί να υπάρξει μια αύξηση, η βελτίωση της απασχόλησης και ένα από τους λόγους γι' αυτό είναι το μείγμα τεχνολογιών που προκύπτει από τον στόχο του 30%. Βλέπουμε σημαντικό ποσοστό υβριδικών ε, ε, οχημάτων που βάζει κανείς στην πρίζα και ε, αυτά τα οχήματα θα έχουν δύο κινητήρες, έναν ηλεκτρικό και έναν ε, κινητήρα εσωτερικής καύσης. Έτσι λοιπόν δεν θα δούμε δραστική μείωση όσον αφορά την απασχόληση. Εάν εξετάσουμε τα στοιχεία της έκθεσης της ΙΤΡΕ, με στόχο 45% το 2025 και 75% το 2030, ο αντίκτυπος ε, θα είναι πολύ ε, πιο δραματικός. Και αν δείτε την πρόταση για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπολογίζονται όλα τα οχήματα χαμηλών εκπομπών και έτσι δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά υβριδικά αυτοκίνητα Ε, δεν θα δούμε λοιπόν σημαντική αύξηση όσον αφορά την απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ομαλή μετάβαση σε οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών που θα επιτρέψει και αρκετό χρόνο για την επανεκπαίδευση των εργαζομένων στην ε, αλυσίδα ε, τροφοδοσίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχουν αρκετές περιφέρειες στην Ευρώπη που εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Νομίζω ότι μπορώ να περιοριστώ σε αυτές τις ε, σύντομες παρατηρήσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ε, μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω συζητήσεις. Ε, νομίζω ότι αύριο μερικοί από εμά θα συναντηθούμε στην Επιτροπή Τραν και Σύντομα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα υποβάλει την γνωμοδότησή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι διατεθειμένη να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και περαιτέρω αναλύσεις, εάν αυτό απαιτείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα να επιστρέψουμε στον συγητή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Έχω κάποια σχόλια για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Κάποιοι φοβούνται ότι πολύ υψηλό στόχο ε, θα δημιουργήσει αναστάτωση στην αυτοκινητοκαινία. Εγώ πιστεύω ότι το αντίθετο ήδη καθυστερεί η Ευρώπη καθώ έχει επικεντρωθεί υπερβολικά στον αδιέξοδο του δίζελ ενώ η Καλιφόρνια, η Κίνα και η Ιαπωνία προωθούν ε, τα οχήματα μηδενικών πομπών. Ε, πρέπει να αναγκαλίσουμε το καινούριο. Η καταστροφή θα έρθει αν συνεχίζει η βιομηχανία να παράγει τα αυτοκίνητα του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος. Και για την κοινωνική προοπτική. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για κοινωνικούς λόγους να καθυστερήσουμε την πράσινη μετάβαση. Όμως, κατά την άποψή μου, αν ε, συνεχίσουμε να ε, καθυστερούμε τη μετάβαση, τότε κατόπιν θα πρέπει να είναι πολύ απότομη η καμπή. Εγώ νομίζω ότι οι επιπτώσεις ε, στην κοινωνία και στην ε, εργασιακή αγορά θα είναι πιο ομαλές αν ξεκινήσουμε τώρα. Κάποιοι μπορεί να ε, ανησυχούν ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ε, νέες δεξιότητες που θα απαιτούνται. Εγώ πιστεύω ότι αν δώσουμε το κατάλληλο πλαίσιο μπορούμε να έχουμε μια πράσινη μετάβαση έτσι ώστε μπορούμε να φτιάξουμε και να εξάγουμε τα αυτοκίνητα του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ να σας ε, υπενθυμίσω ή να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών είναι στις 26 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι 26 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, πρόθεση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, οδικών μεταφορών. Ο εισηγητής είναι ο κύριος ε, Τούρμες και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να παρουσιάσει την εκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Οι δημόσιες ε, προμήθειες από τις κυβερνήσεις αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση όταν μιλάμε για τις δημόσιες προμήθειες για τα οχήματα αν ε, η τοπική αυτοδιοίκηση ή ένα σύνολο ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, κάνει ένα διαγωνισμό για τη συλλογή, την αποκομιδή των απορριμμάτων μπορεί να αποφασίσει για το είδος των οχημάτων. Δηλαδή αυτό είναι πιο ευρύ από τα αυτοκίνητα ή τα οχήματα που η τοπική αυτοδιοίκηση θα αγοράσει η κυβέρνηση, αλλά μιλάμε και για τις δημόσιες προμήθειες υπηρεσιών που συνοδεύουν τα οχήματα αυτά η Κομισιόν είχε μια παρουσίαση μια φυστάμενη οδηγία ήταν τόσο δύναμη που δεν λειτουργούσε στην πραγματικότητα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια αναθεώρηση και νομίζω ότι είναι καλό που παρουσιάζει η Κομισιόν αυτή την αναθεώρηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια σημεία. Κάποιοι λέτε τεχνολογική ουδετερότητα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι σε ένα κόσμο κλιματικών αλλαγών <laughs> αυτό είναι ανοησία. Έχετε ένα πλανήτη όπου έχουμε ρήπανση ε, από άνθρακα, πρέπει να κλείσουν ε, η παραγωγή του λιγνίτη και των ορυκτών καυσίμων. Έχουμε λοιπόν μία σειρά τεχνολογιών που είναι επιλέξιμες και έχουν διάφορους βαθμούς αποδοτικότητας. Έτσι λοιπόν είναι σχετικά προφανές, αν το δείτε εις βάθος το θέμα, ότι τις επόμενες δεκαετίες θα έχουμε ηλεκτρικά οχήματα και κάποια υβριδικά. Και πιθανότητα ε, η παραγωγή υβριδικών τι σημαίνει ηλεκτρικό υδρογόνο. Αυτή είναι μια πιθανή επιλογή. Και στη συνέχεια το ένα θέμα αφορά τη ρήπανση, αλλά έχουμε να δούμε και το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής και σας δώσω ένα αριθμητικό στοιχείο και μπορώ να σας πω τρακούνισε την Κομισιόν στην Κίνα. Σήμερα έχουμε 400.000 ηλεκτρικά λεωφορεία. Πόσα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουμε στην Ευρώπη? Ούτε καν 2.000. ούτε καν 2.000. Δεν ε, υπάρχει καμία μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία παραγωγής λεωφορείων που να έχει εναγκαλίσει την παραγωγή ηλεκτρικών λεωφορείων ενώ στην Κίνα έχουμε 5-10 εταιρείε που έχουν παράξει ήδη χιλιάδες λεωφορεία ναι, λοιπόν η βιομηχανική μας πολιτική θέλουμε να επιβιώσει, πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και τι θέλω να κάνω με τις ε, δημόσιες προμήθειες, με τη βοήθειά σας, είναι να δημιουργήσω ε, μία αγορά για ηλεκτρικά υβριδικά οχήματα και για οχήματα με υδρογόνο που θα οδηγήσει στην παραγωγή μπαταριών επόμενης γενιάς. Γιατί με την μπαταρία είναι πολύ εύκολο. Ζητάς από μια εταιρεία, ρωτάς μια εταιρεία σήμερα που μπορώ να αγοράσω τις πιο φθηνές μπαταρίες, η απάντηση είναι όχι στην Ευρώπη. Η LG από την Νοτιοκορέα ή από την Κίνα ή η Panasonic από την Ιαπωνία. Το έχουμε συζητήσει αυτό με την Κομισιόν και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος να επανέλθει η Ευρώπη στο παιχνίδι είναι να μεταβεί στην πράσινη μπαταρία 100% ανακυκλώσιμη που σημαίνει εξσχεδιασμού ανακυκλώσιμη, δηλαδή πρέπει να σχεδιάσει την μπαταρία έτσι ώστε εξ αρχή ξέρει ότι στη συνέχεια μπορεί να την αποσυναρμολογήσει και να την ανακυκλώσει. Δεύτερον, ε, τα ε, ε, φάσματα της μπαταρίας θα πρέπει να τρέχουν με 100% ε, ενέργεια από ενενέσιμες πηγές και το τρίτο θέμα είναι οι πηγές. Το μπορεί να γίνει εν μέρει στην Ευρώπη και μπορούμε να έχουμε και μια πρωτοβουλία για φόρο εξόριξη. Έτσι λοιπόν εδώ δεν μιλώ μόνο για την αγορά ενός ποσοστού ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά το συνδέω αυτό και με τις μπαταρίες που θα υπάρχουν στα αυτοκίνητα αυτά. Και έχω αναφέρει κάποια νούμερα που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Το σημαντικό είναι ότι η Κομισιόν δεν έχει νούμερα για το 2020. Η δική μου ανάλυση είναι ότι τώρα ήρθε η στιγμή που θα νικήσουμε ή θα χάσουμε. Υπάρχει μια αγορά το 2020, θα έπρεπε να υπάρχει μια αγορά που να δημιουργήσει μια αγορά αριστεία στην Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για μια υποχρέωση που θα επιβληθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και μπορώ να σας πω η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τιμή να συμμετέχει στο παιχνίδι, αλλά υπάρχουν και χρήματα βέβαια. Έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρομαι στα χρήματα από το ΕΦΣΥ, ε, στο Μηχανισμό Συνδέοντας στην Ευρώπη κτλ. Υπάρχουν χρήματα λοιπόν για να βοηθήσουμε να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Επίσης, μην σκέφτεστε ότι μπορείτε να απορριπάνετε πολύ γρήγορα τις πόλεις, μόνο αν επικεντρωθούτε ε, σε το καινούριο. Έχουμε ε, 253 πόλεις στην Ευρώπη που δεν σέβονται τα πρότυπα σε ό,τι αφορά τη ρήπαση του ατμοσφαιρικού αέρα. Για αυτές τις ε, πόλεις, για αυτήν την κατηγορία προτείνω ένα ειδικό πρόγραμμα μετασκευής που ε, προσανατολίζεται πολύ περισσότερο στον ηλεκτρισμό γιατί σε δύο-τρία χρόνια πρέπει να παράξει αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ε, μετασκευή, επίσης ε, να έχουμε στα ίδια υβριδικά λεωφορεία περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το πώς θα φέρουμε γρήγορα αποτελέσματα σε αυτές 350 πόλεις στην Ευρώπη που παραβιάζουν την παραβιακή νομοθεσία. Αυτή είναι μια σύνοψη των προτασιών μου. Ευχαριστώ κύριε Τούρμες. Και τώρα για το ΕΛΚ. Ο κύριος ε, Γκάμπους, δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Τούρμες για τη δουλειά του έως τώρα για το ζήτημα αυτό και για το γεγονός ότι θα τροπολογίες ε, ε, στην πρότασή του ε, είμαστε μάλλον αρκετά μακριά από την άποψή του αλλά θα, πραγματικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να φτάσουμε σε συνένεση, σε ένα ισορροπημένο κείμενο με ευρεία υποστήριξη. με βέβαια ότι ε, και, και οι τροπολογίες των λοιπόν ομάδων θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο σταθερό και κάποιοι στόχοι σαφείς, προκαθορισμένοι και εφαρμόσιμοι, πραγματοποιήσιμοι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τι διεθνεί τη δεσμεύσει, ιδιαίτερα ε, τη Συμφωνία των Παρισίων. Όμω δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι αυτοί οι στόχοι, του οποίου δεν μπορούμε να παρνηθούμε βέβαια, δεν μπορούν να πάνε ενάντια σε μια διαδικασία ε, ε, επαναβιομηχανοποίηση τη Ευρώπη. Μια βιομηχανία που πρέπει να είναι ανταγωνιστική, καινοτόμα και να δημιουργεί θέσει εργασία ε, υψηλών δεξιοτήτων ή δυνατών. Σε αυτή την προσπάθεια επαναβιομηχανοποίησης ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι ε, για να μειωθεί οι εκπομπές ε, και η ρήπανση ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωράει η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η έρευνα και τεχνολογία. πρέπει να προχωρήσουμε επίσης στην διαδικασία ε, εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τι δημόσιε προμήθειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε μια αγορά υψηλού επίπεδου για τα λεωφορεία, τα φορτηγά, ε, τον εξοπλισμό. Ε, αν δεν έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η καινοτομία και οι επενδύσει στην ε, καθαρή. Ε, ε, στι καθαρέ μεταφορέ δεν θα είναι ανταγωνιστική ευρωπαϊκά. Ε, παγκοσμίω μάλλον. Οποιαδήποτε πολιτική δεν μα επιτρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκοσμίω ε, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ε, πρέπει να είναι σαφές για μας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία, ε, την ευρωπαϊκή από τον αθέμητο ανταγωνισμό τρίτων χωρών ε, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες μεταξύ άλλων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει πολλά μέτωπα, έχει προσθέσει ακόμα μερικά μέτωπα ο εισηγητής για κάποια από αυτά, με κάποια από αυτά συμφωνούμε, με κάποια άλλα διαφωνούμε. Οι τροπολογίες μας θα ακολουθήσουν τη φιλοσοφία ε, της παρέμβασης που μόλις ακούσατε. Πρόθεσή μας είναι πάντως ε, η, η ορθή λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της βιομηχανίας της, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ο συντονισμός, ε, η, η διατήρηση μάλλον του κράτους δικαίου, όπου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική η οικονομία μας, και ο σεβασμός ε, των διεθνών δεσμεύσεων μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε πόσο μας να τα συγκεράσουμε. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες αυτού του Κοινοβουλίου υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και τώρα ο κύριος Κορουμπάση, Κορουμπάσεφ συγγνώμη, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τις υποδομές που χρειαζόμαστε διότι έχουμε περίπου 120.000 ε, σημεία Φόρτωση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε 6-7 φορές περισσότερα. Χωρίς αυτή την υποδομή ε, δεν μπορούμε ε, να επιβάλλουμε στους παραγωγούς να επιτύχουν μόνοι τους τους στόχους. Χρειαζόμαστε επιπλέον χρηματοδότηση λοιπόν και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες και σε ό,τι αφορά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτό έχει να κάνει και με το τις μεταφορές επιβατών αλλά ε, και για ε, τα άλλα οχήματα ε, τις δημόσιες μεταφορές αυτό επηρεάζει τον προπολογισμό και τον δημοτικό σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο ο μηχανισμός του Connecting Europe είναι ένα χρήσιμο εργαλείο χρηματοδότηση τέτοιου project για να καλύψουμε ε, τα σημεία, τα κενά που υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίση μπορεί να αποτελέσει πηγή χρηματοδότηση. Στο πολιτισμό, μας νομικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτά τα στοιχεία στις διατάξεις του και κάτι άλλο. Το σύνολο του κύκλου ζωής ε, ενός οχήματος ε, θα πρέπει να αξιολογηθεί ε, όχι μόνο σε επίπεδο εκπομπών, αλλά και το τι εκπέμπουμε για να το παράγουμε και για να το ανακυκλώσουμε αυτό το λεωφορείο. Αυτό θα μας δώσει μια πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διεξίου του άνθρακα για το σύνολο του κύκλου ζωής, επαναλαμβάνω, ενός ε, λεωφορείου, ενός οχήματος. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε παραγωγές που θα μας επιτρέψουν να παράγουμε προϊόντα με χαμηλότερες εκπομπές και να μπορούν να κυκλοθούν και πιο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Στοζανόσκη τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ε, δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβω αυτά που είπα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο της έκθεσης. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είτε μιλάμε για πολύ φιλόδοξη πρόταση, είτε για τον τρόπο να βρούμε ε, την καλύτερη τεχνολογική λύση. Μια διευκρίνηση όμως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Στις ε, δημόσιες μεταφορές, ε, στις μαζικές μεταφορές υπάρχουν ε, συστήματα μηδενικών εκπομπών. Για παράδειγμα τα τρένα είναι ηλεκτρικά. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί στις αστικές περιοχές και υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τα συστήματα συσσωρευτών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις μπαταρίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι έχουν μεγάλο χρόνο φόρτισης. Δεν μας παίρνει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τέτοια συστήματα και τα λέω αυτά ως πρώην δήμαρχος μεγάλης ε, βιομηχανικής πόλης όπου είχαμε ξεκινήσει τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είμαι πεπισμένο ότι υπάρχει επαρκέ τεχνολογικό δυναμικό για ώστε να αναπτυχθεί νέο σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή όμως οι μπαταρίες που έχουμε στη διάθεσή μας αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις πόλεις, ούτε υπάρχει σταθμός φόρτισης σε κάθε γωνία. Εάν κάθε λεωφορείο πρέπει μετά από κάθε ώρα χρήση ε, να πρέπει να φορτίζει δύο ώρες, ε, αυτό δεν έχει νόημα, διότι χρειαζόμαστε τα δεκαπλάσια οχήματα τότε. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή, γι' αυτό θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Δεν ε, θα πρέπει όμως να προδικάσουμε τις εξελίξεις διότι μπορεί κάτι να φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι η μοναδική λύση, μπορεί όμως να μην είναι. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις διάφορες λύσεις ε, θα πρέπει να τις εξετάσουμε στο πλαίσιο των πόλεων. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των φιλοδοξιών, φιλοδοξιών μας. Ε, αυτά από μένα προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τόσενόφσκι. Από την άλλη η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά τον ε, εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Συμφωνώ ε, σε κάποια από τα θέματα, σε άλλα όχι. Θα ξεκινήσω από αυτά στα οποία συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος ε, να πούμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα με τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων. και ε, όπως λέει και η πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει να εξετάσουμε το συνολικό κύκλο ζωής διότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο ε, να δούμε τι, τι εκπομπές ε, εκπέμπει το όχημα, θα πρέπει να δούμε και την διαδικασία παραγωγής και παροπλισμού. Όσον αφορά την ηλεκτροκινητικότητα, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε τεχνολογικά ουδέτεροι. Έχουμε κάποιες ε, λύσεις ε, στην Ευρώπη όπου θα μπορέσουμε να αναλάβουμε και ηγετική θέση. Έχουμε για παράδειγμα προηγμένα βιοκαύσιμα. Υπάρχουν ε, συνθετικά καύσιμα τα οποία μπορεί να δούμε στο μέλλον. Η Σκανδιναβία ποντάρει περισσότερο στο αέριο από ό,τι στην ηλεκτροκινητικότητα. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για τα εναλλακτικά καύσιμα, την οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε όχι μόνο στον τομέα της ηλεκτροκινητικότητας, ε, αλλά και ε, σε άλλους τομείς, ε, όπως είναι το υδρογόνο κλπ. Τίθεται και το θέμα του τι άλλο θα προταθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατικών Επενδύσεων κλπ. της διευκόλυνσης ε, συνδέοντας σε την Ευρώπη. Αυτά που έχουμε στο πλαίσιο του Euro 6 δεν είναι πολύ ε, άσχημα. Ε, και επίση θα πρέπει να εξετάσουμε ότι ο μεταξοπλισμός μπορεί να οδηγήσει ε, στην πλήρη απουσία μεταφορών ε, στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας και γι' αυτό θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σορίνιο. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Σε αυτές τις δύο τελευταίες γνωμοδοτήσεις προσπαθήσαμε να έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση για το μέλλον της κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα είναι ότι έχει επαναληφθεί πολλές φορές ε, ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ηγετική θέση ε, όμως ε, αυτό δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Εμείς θα πρέπει βέβαια να είμαστε φιλόδοξοι Γι' αυτό συμφωνώ με την εξή προοπτική. Αφενός ε, θα πρέπει να έχουμε μικρά βήματα στην ε, προσαρμογή των σημερινών μοντέλων, αλλά θα πρέπει να στοχευσούμε και στην ε, νέα τεχνολογική γενιά και στις πράσινες μπατερίες και να έχουμε και ένα δίκτυο φόρτισης νέας γενιάς που να είναι τεχνολογίας εχμής. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τάσεις οργάνωσης της κοινωνίας συνδυάζοντας την ενέργεια και την πληροφόρηση. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο θα παρουσιάσει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Η προτεραιότητα για να έχουμε καθαρή κινητικότητα και των υποδομών φόρτισης θα πρέπει να ε, είναι ξεκάθαρες σε αυτό το πλαίσιο και θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι στον ορίζοντα 2020 θα πρέπει ε, να θέσουμε ε, τους μηχανισμούς πρόθεσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και το κατάλληλο δίκτυο φόρτισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζωρίνη. Κύριος Νίκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι μου αρέσει η έκθεση επί της αρχής γιατί θίγει μια προοπτική που ε, τη συζητούμε εδώ και καιρός. Ό,τι αφορά τώρα τα μέσα μεταφοράς. Τα μέσα μεταφοράς ε, πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όμως ε, δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ακούσαμε ότι η Κίνα ε, αγοράζει λεωφορεία υβριδικά, όμως κανείς δεν ξέρει να δώσει πληροφορίες στην Ευρώπη πώς ε, μπορεί να αγοράσει αυτά τα λεωφορεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά τα λέω και προς εκπροσώπους της Δεύτερον, πήγα στο Σαν Φρανσίσκο πριν δύο εβδομάδες, στο Σαν Φρανσίσκο ε, βλέπετε ε, καινούριε ε, μεταφορές, έχουμε λεωφορεία που δεν παράγουν εκπομπές, τραμ. Όμως πάνω από 90 του στόλου στο Σαν Φρανσίσκο είναι εντελώς καινούριο. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Δεύτερον, ε, σε ό,τι φορά ε, τα βαριά εμπορικά οχήματα, στα βαριά δεν ξέρω ούτε μία ε, περίπτωση ενός οχήματος που να ε, λειτουργεί με ηλεκτρική μπαταρία. Για τα ελαφρά οχήματα όμως θα μπορούσαμε να έχουμε μπαταρίες που είναι διαθέσιμες τώρα και να έχουμε ελαφρά εμπορικά οχήματα. Ε, το θέλω να πω δύο πράγματα να σκεφτεί ο εισηγητής. Καταρχήν, το βάρος της μπαταρίας ε, σημαίνει ότι ε, ουσιαστικά αυξάνεται και το βάρος του οχήματος πάνω από το επιτρεπόμενο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το θέμα και θα πρέπει να υπολογιστεί η κατηγορία των οχημάτων ανά βάρος. Και το δεύτερο είναι ε, το θέμα που ε, ε, το χάρη ε, το θέμα της προβλεψιμότητας χρειάζονται πριν το σχάρι 7 χρόνια ε, για να μπορεί να σχεδιαστεί ένα νέο όχημα και να μπορεί να τεθεί προς πώληση. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια προβλεψιμότητα για όλους αυτούς ε, τους παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ το θέμα αυτό της προβλεψιμότητας επίσης να ληφθεί υπόψη για να μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη παραγωγή που να μπορεί να τεθεί ε, σε εφαρμογή. Επίσης, ε, νομίζω ότι για ορισμένες ε, χώρες δίνονται πάρα πολλά κίνητρα. Αν δούμε τι γίνεται στη Ρουμανία, 75% μέχρι το 2050 ή μέχρι το 2030 για τεχνολογίες μηδενών εκτών είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος αυτός για τη χώρα μου. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα τεχνολογικά βήματα που θα μας οδηγήσουν σε ένα τέτοιο ποσοστό. Ίσως ε, να μην είναι καλά τα παραρτήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραρτήματα με τις υποχρεώσεις για κάθε κράτος μέλος και για τα βαρέα οχήματα. Στα βαρέα οχήματα είμαι ακόμη πιο σκεπτικός αν υπάρχει και μια μοναδική περίπτωση ε, παγκοσμίω να έχουμε ένα φορτηγό ε, που ε, να λειτουργεί με ε, ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, όλοι στην Ρουμανία θα αναρωτηθούν τι έχετε κατά νου αν παρουσιάσετε τέτοια ποσοστά. Επίσης, δεν πρέπει να υιοθετήσουμε μια πρόταση που να μην είναι μη ρεαλιστική. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, εμπειρογνώμονες στον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για την Κομισιόν ο κύριος Σοντομπολίνο. Ευχαριστώ που δίνετε στην Κομισιόν την ευκαιρία να κάνει κάποια σχόλια και να δώσει κάποιες εξηγήσει. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση αυτή που ενισχύει το επίπεδο φιλοδοξίας της Κομισιόν. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω μία πτυχή που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και σε σχέση με τα τελευταία σχόλια για τη διαθεσιμότητα των ε, ηλεκτροκινούμενων φορτηγών, η πρόταση της Κομισιόν. Ε, εξετάζει τα καθαρά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών κουμπών. Δεν αφορά μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή προς αποσαφήνιση, πιστεύω. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, δηλαδή τα αυτοκίνητα και τα βαν, η πρόταση λέει ότι τα κατόβλια των εκπομπών για το 2025 που τίθενται στα 25 και στα 40 γραμμάρια, αυτό θα είναι ε, τα πιο αποτελεσματικά φορτιζόμενα ευρυδικά που έχουμε και θα έχουμε μηδενικό, στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2030. Σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα, η πρόταση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή είναι να συμπεριληφθεί ο ηλεκτρισμός, το υδρογόνο και το φυσικό αέριο εμείς ζητούμε να μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτά όταν θα έχουμε τα πρότυπα για τα βαρέα οχήματα. Τώρα, έχει προτείνει ο εισηγητής διαφορετικά κατόφλια ήδη ε, με κατόφλια εκπομπών για τα βαρέα οχήματα. Είναι λοιπόν πιο συνεκτική η πρότασή σας, αν θέλετε. Όμως, ε, ε, επίσης, δεν έχουμε μόνο ε, το όριο του 2025. Όταν δηλαδή βλέπουμε το στόχο του 2025 δεν έχουμε μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για μετέπειτα στάδια έχουμε μηδενικέ εκπομπές με οποιαδήποτε τεχνολογία είναι διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή για την επίτευξη του στόχου. Άκουσα πολλά σχόλια για το θέμα του κύκλου της ζωής. Φυσικά αυτά τα παίρνουμε πολύ σοβαρά και εξετάζουμε τις διάφορες επιλογές. Όμως ό,τι αφορά το θέμα τη συνεκτικότητας με άλλες νομοθεσίες και να αποφύγουμε τα προβλήματα με την ε, κατανομή, ε, λαμβάνοντα υπόψη και τις ε, άλλες νομοθετικές προτάσεις, θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή που σχετίζεται με τις δημόσιες συμβάσεις των αυτοκινήτων είναι η καλύτερη οδός με τις περιορισμούς που έχει. Όμως αυτή τη στιγμή αυτή είναι η μόνη λύση που βλέπουμε για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πτυχή των οχημάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύκλο της ζωής ε, και ε, το θέμα από τη δεξαμενή ε, στον τροχό και τη διαθεσιμότητα των υποδομών, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι προτάσεις είναι μέρος ενός πακέτου. Δεν θα λύσουμε τα πάντα με την πρόταση αυτή. Έχουμε μία οδηγία, όπως ξέρετε, για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων και έχουμε δράσει από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά και για την προώθηση των τεχνολογιών ε, για τις μπαταρίες και τις πιο αηφόρες μπαταρίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις μπαταρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση έχουμε την οδηγία για τις ανάσχημες πηγές ενέργειας, όπου εξετάζουμε το θέμα ε, του από πού πηγάζει η ενέργεια για διάφορου τομεί και για τις μεταφορές. Αυτή η πρόταση αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες, τις δημόσιες συμβάσεις οχημάτων. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τις συγκεκριμένε πτυχέ που σχετίζονται με τα οχήματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητής ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ συναδέλφους για τα πολύ ψυχμηρά σχόλια, για τις υποδομές. Έχετε δίκιο, κύριε Κορομπάτσεφ, αλλά εδώ μιλάμε για τους νέους τόλους. Μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Εδώ μιλάμε για λεωφορεία. Πρέπει απλώς κάποιος στον τεπό του να έχει μια υποδομή φόρτισης και σε κάποια στρατηγικά σημεία ακόμα. Δηλαδή το πρόβλημα της υποδομής, το οποίο συνδέεται με το γεγονό ότι η Κομισιόν δεν τολμάει να κάνει μια πλήρη αναθεώρηση των υπάρχοντων εναλλακτικών και τη σχετική οδηγία, ε, δεν, δεν υπάρχει το πρόβλημα εδώ με τι υποδομέ Εδώ μπορούμε να πάμε γρήγορα. Εάν μια πόλη αγοράσει ηλεκτρικά λεωφορεία και έχει πρόσβαση στα κονδύλια τα ευρωπαϊκά πρέπει να είναι επιλέξιμη και για τις, τους σταθμούς φόρτισης και στις συζητήσεις που είχαμε στις μεγάλες πόλεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια πρόκληση και για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, διότι έχουμε πολλούς μηχανικούς, μεγάλη πραγματονομοσύνη μηχανικών, που θα πρέπει να περάσουν τώρα σε μια πραγματονομοσύνη ηλεκτρική. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές για τα pentographs τώρα. Όταν μιλάω με τις εταιρείε λοφορείων, μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, διότι είναι πολλές εταιρείε που πολλούν pentographs, αλλά το λογισμικό τους ε, δεν επιτρέπουν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα λεωφορεία. Ε, όλη αυτή η συζήτηση τώρα για τον κύκλο ζωής. Θα πρέπει να υπάρξουν λεπτομερείς αναλύσεις. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, ποια θα είναι σε πέντε χρόνια. Ιδάλλως, το Dieselgate, ε, ή μάλλον αυτοί που κάνουν Dieselgate θα μας κατηγορούν ότι δεν είναι καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τα δικά τους. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Όμω χρειαζόμαστε στοιχεία για να το αποδείξουμε. Και ο μόνος μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα, ε, τα φορτηγά, ε, σημαντικό αυτό. Με την eBay, με το Amazon, ε, έχουμε όλο και πιο πολλά φορτηγάκια. Λιγότερα φορτηγά μεγάλα δηλαδή και πιο πολλά μικρά βανάκια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις πόλεις και για τη, και για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη της ατμόσφαιρας. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και εκεί. Εκεί μπορούμε να πάμε γρήγορα και για τα υβριδικά, ηλεκτρικά. Τώρα, πράσινη μηχανική. Υπάρχει το θέμα τη χορύπανση. Μεγάλο πρόβλημα τη πόλη μα. Φανταστείτε με αυτή την νομοθεσία να έχουμε ένα σημαντικό αριθμό μεγάλων πόλεων στις επόμενες, ε, στις επόμενες συμβάσεις να ε, επιβάλλουν ηλεκτρικούς κινητήρες. Αυτό θα μειώσει δραματικά την ηχορύπανση. Και χωρίς το, μια αγορά που να το σπρώξει αυτό δεν πρόκειται να καταφέρουμε. Λοιπόν, οι δημόσιες προμήθειες μπορούν πραγματικά να δώσουν μια όθηση. Εφόσον γίνουν σωστά. Βεβαίω υπάρχουν βιοκαύσιμα, βεβαίω υπάρχει το αέριο. Αλλά δεν, έχετε, δεν, έχετε, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει επακριβώ η Συμφωνία των Παρισιών. Μηδέν το 2050. Ένα φορτηγό έχει διάρκεια ζωή 25, 30, 40 χρόνια. Εάν αφήσετε λοιπόν ένα αέριο το 2030 για ένα φορτηγό, ένα φορτηγό αερίου, θα είναι εκεί και το 2050 αυτό το φορτηγό. Με το Παρίσι θα πρέπει να σκεφτούμε προς τα πίσω, πολύ πριν. Πότε θα πρέπει αυτή η τεχνολογία ε, να κλείσει τον κύκλο ζωής της. Και το άλλο επιχείρημα κατά των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιείται εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε βιοκαύσιμα για τα αεροπλάνα. Θα έχουμε κάποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι χρηματοδοτούμε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Rolls Royce, στην Airbus, για να παράξουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά για 30, 60 ε, επιβάτες. Για τα μεγάλα όμως οχήματα, ε, αυτοκίνητα ε, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Η μόνη εναλλακτική στην κεροζίνη είναι τα βιοκάσιμα. Τα βιοκάσιμα όμως είναι περιορισμένα ε, σε, σε ποσότητα. Το συζητάμε και με τον κύριο Χάνκελ που μας υποστήριξε να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα. Τα βιοκαύσιμα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έχουμε ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε ε, υβριδικά για τα οχήματα, τα φορτηγά, τα επιβατηγά, αλλά όχι για τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη. Αυτό είναι άλλο ένα δίλημα που πρέπει να, να απαντήσουμε. Και όταν κάποιος στη Ρουμανία σε ρωτάει πού να αγοράσω το πράσινο λεωφορείο, Υπάρχει μια πλατφόρμα πράσινων λεωφορείων. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία χρηματοδοτεί ο κοινωνικό προπολογισμό που διάφορε πόλει αυτή τη στιγμή από κοινού εμπειρογνώμονε ορίζουν ε, πώ ε, γίνεται ο διακονισμό σχετικό και έχουμε και σχετικέ εμπειρίε. Πρέπει όμω η Κομισιόν να μα δώσει μεγαλύτερη τεχνική συνδρομή, διότι χάνουμε, χάνουμε χρόνο με λάθη που κάνουμε. Διότι δεν έχουμε τις καλύτερες ε, διαθέσιμες πληροφορίες στη διάθεσή μας και για την Ήπεθρο. Στην Ήπεθρο έχουμε πέντε λεωφορεία. Εάν αγοράσουν δύο καινούρια λεωφορεία, έχουν φτάσει σχεδόν στο 50% ήδη. Μόνο όταν αγοράζει κανείς κάτι καινούριο, σας βοηθούμε και σας ζητούμε να αγοράσετε νέας γενιάς ε, όχημα. Δεν σας, δεν σας υποχρεώνουμε να, να πουλήσετε νωρίτερα ε, το λεωφορείο σας, να το αγοράσετε νωρίτερα το καινούριο. Στις 400 πόλεις όπου ε, υπάρχει θέμα ε, αθμοσφαιρικής ρήπανσης, προτείνω ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο, στη νέα αγορά. Διότι η νέα αγορά είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλα τα λεωφορεία του Βερολίνου. Κοστίζει πάρα πολύ. Κάποια λεωφορεία λοιπόν θα πρέπει να επανέλθουν και να ε, τροποποιηθούν. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία να μπορούν να κάνουν και εκεί αυτό. Έχει και δίκιο ο κύριος Γιούνκερ. Δεν θέλουμε εδώ ένα χάσμα Ανατολής Δύσης. Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα σε, σε, σε επίπεδο πόλης σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, να τους βοηθήσουμε. Λοιπόν, ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε μια όθηση στους Ευρωπαίους στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Τούρμες να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την υποβληθούν τροπολογίες είναι η 30 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. 12 το Κυρίε και κύριοι, έχουμε ακόμα δύο σημαντικούς φάκελους. Θα ήθελα να περάσουμε στον επόμενο. Ενημέρωση για τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσει. Η οδηγία για τις πηγές ενέργειας. Ο Χωσέ Μπλάνκο Λόπεθ είναι ο εισηγητής, όμως δεν βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ε, ζήτησε λοιπόν από μένα να συνοψίσω την κατάσταση, το που βρισκόμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή και θα το κάνω ε, πολύ γρήγορα. Ο δεύτερος τρίλογος για, τις, για τα ανανεώσιμα έλαβε χώρα την Τρίτη ε, 27 Μαρτίου. Οι, σχέσεις, οι θέσεις μάλλον των ε, συνομοθετών αποκλίνουν σημαντικά για πολύ σημαντικά ζητήματα μάλιστα σε ό,τι αφορά τον συνολικό στόχο για την κατανομή των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και το ποσοστό μάλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, υπάρχει ακόμα στο 27% από το Συμβούλιο. Είχαμε στήσει να αυξηθεί η φιλοδοξία στην, ε, μετά την σύνοδο των Υπουργών στη Σόφια την περσμένη εβδομάδα δεν σημειώθηκε όμως πρόοδος έγινε και μια απόπειρα να σημειωθεί πρόοδος επί βουλγαρικής προεδρίας έγιναν κάποιες τεχνικές συναντήσεις με τον τελευταίο τρίλογο και προβλέπονται και άλλες συνεδριάσεις πριν τον επόμενο στις 17 Μαΐου. Ε, η προσωρινή συμφωνία έχει επιτευχθεί για μια σειρά από άστρα οι μεταφορές, η Επιτροπή Μεταφορών, στην Επιτροπή Μεταφορών μάλλον γίνεται συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο, ο εισηγητής θέλει να υπογραμμίσει εδώ ότι υπάρχει έλλειψη φιλοδοξίας στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αύξηση του ποσοστού, του μεριδίου των ε, ανανεώσιμων στον τομέα των μεταφορών. Ελπίζουμε στο νέο τρίλογο το Μάιο, στι 17 Μαΐου αλλά και στις 29 Μαΐου, δύο, δύο συνεδριάσεις, η Προεδρία θα μπορέσει να λάβει μια ευρία εντολή για να διαπραγματευτεί και να υπάρξουν πραγματικοί συμβιβασμοί για όλες τις σημαντικές διατάξεις αυτού του φάκελου. Και ο εισηγητής επίσης ε, ευχαριστεί τους και όλους εισηγητές και τις ομάδες τους για την εξαιρετική συνεργασία. Τώρα, ε, από το ΕΛΚ ο κύριος Κέλλη δεν είναι εδώ. Α, κύριε Τούρμες, θέλετε να μας πείτε από αυτού. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Ναι, ναι, έχω πολλές ε, ταυτότητες σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Μπλάνκο περιέγραψε πολύ καλά την κατάσταση. Έχουμε μια σαφή θέση εμείς στο Κοινοβούλιο και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια θέση του Συμβουλίου που είναι πολύ μακριά από τη δική μας. Το πρόβλημα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση είναι ότι εφόσον το Συμβούλιο δεν κάνει καμία κίνηση, δεν έχει νόημα, δεν προχωράμε. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να ε, εξετάσουμε τα εύκολα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουμε τα χατιά μας ε, για τα πιο βασικά. Η φιλοδοξία που, του, του, όλης πρότασης, το πώς θα κατανείμουμε τους στόχους και των μελών, μεταφορές, ε, θέρμανση. Ε, ο κύριος Μπλάνκο το προχωράει σωστά το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία. Ε, για την συνδρομή, την πολύτιμη συνδρομή υψηλού επίπεδου που μας παρέχει. Μάλιστα. Ε, εγώ είμαι σκιώδης συγκητής σε ό,τι αφορά την ECR να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια ε, για τις δικές μου εντυπώσεις. πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν εξαιρετικά αργά. Δεν είμαι βέβαιος για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε επί βουλγαρικής προεδρίας. όπως ήδη υπόθηκε, όπως είπε ο κύριος Μπλάνκο, ε, υπάρχουν ζητήματα που εκκρεμούν τα οποία είναι εξαιρετικά αφιλεγόμενα σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση τομέα των μεταφορών θα χρειαστούν ε, πιο προχωρημένα βιοκαύσιμα ε, και συμβατικά κάποιοι θέλουν να υπάρξει όμως απόλυτη κατάργηση των βιοκαυσίμων σταδιακά η παραγωγή όμως βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς πρέπει να συμφωνηθεί και με τους εμπορικούς εταίρους μας. Ε, και δεν καταλαβαίνω αυτό με την, ε, την ηλεκτρική ε, μετάβαση. Πρέπει να είμαστε πιο ουδέτεροι. Εγώ στην αρχές Μαΐου θα δοκιμάσω για μία εβδομάδα ένα αυτοκίνητο υδρογόνου. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για την εμπειρία μου θα σας ενημερώσω σχετικά. Πρέπει να πω βέβαια ότι βλέπω ότι υπάρχουν καλές προσφορές μόνο από Ιάπωνες ε, κατασκευαστές και αυτό με σώκαρε κάπως. Τον Ιούνιο του 2017 η Παγκόσμια Τράπεζα ε, ε, παρουσίασε μια έκθεση για το πέρασμα προς την καθαρή ενέργεια αναφέρει ότι είναι πιο τα συστήματα παροχών βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα για τις μπαταρίες και τις τουρμπίνες θα θα εξαρτώμεθα από εισαγωγές από χώρες με μικρή παραγωγικότητα ε, και αυτό θα πρέπει να ε, θα γίνουν ουσιαστικά ε, αποθήκες όπως στο Κονγκό, στη Βολιβία για το λίθιο. εδώ σας συστήνω ένα κείμενο που δημοσίευσε η κυρία Οσάλιβαν από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για τα γεωπολιτική των ανανεώσιμων αυτή η ιδέα ότι οι ανώσιμες πηγές ενέργειας θα μας καταστήσουν πιο ε, ανεξάρτητους ε, πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι που, αυτό ισχύουν, που ισχύουν και για τη βιοπικιλότητα. Όσο μεγαλύτερη ποικιλομορφία υπάρχει τόσο πιο ανθεκτικός είναι κάποιος. Τέλος για το θέμα ε, υπάρχουν εδώ, υπάρχει ιδεολογική, δογματική προσέγγιση. Εμείς δεν συμφωνούμε με τον συμβασμό ALDE, ε, EPP και S&D και για το Φινικέλεο, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση. Εγώ συνάντησα τον Κολομβιανό Υπουργό Γεωργίας και την αντιπροσωπεία του σήμερα το πρωί και θα ήταν καλό να τον είχατε δει όλοι, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση. Επικεντρωθήκαμε στο ρόλο της, του τομέα της γεωργίας και της παραγωγής φινικελαίου ιδιαίτερα ε, στην διαδικασία ειρήνευσης και το πώς μπορεί αυτός ο τομέας να ε, επανεντάξει μαχητές και πολεμιστές ε, στον τομέα της γεωργίας στις ευαίσθητες περιοχές της Κολομβίας, τους μαχητές της ΦΑΡΚ. Ε, έγινε αναφορά στο ότι πρέπει οι μικροί γεωργοί να έχουν περισσότερες δυνατότητες, ιδιαίτερα ε, στην Κολομβία. Πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση όταν μιλάμε για φινικέλαιο, διότι ο τρόπος με τον οποίο παράγεται, το έδαφος επί το οποίο παράγεται, αν αυτό γίνεται σε ένα δάσο ή σε μια ζούγκλα, αν πρέπει να κοπούν δέντρα, ε, είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Πρέπει να γίνει διαφοροποίηση. Λυπάμαι που άκουσα ότι αυτή η ομάδα δεν μπορούσε καν να συναντηθεί από κάποιους εισηγητές αυτή η ομάδα του Υπουργού. Εγώ συναντώ τους πάντες, ε, την Greenpeace, ε, την WWF, ε, την BirdLife, όποιον θέλετε. Γιατί οι πράσινοι και κάποιοι άλλοι, ή κάποιοι σοσιαλιστές σε αυτό το κοινοβούλιο αρνούνται να μιλήσουν με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Ελπίζω να είναι εξίσου ανοιχτοί οι συνάδελφοι, να είμαστε ανοιχτοί απέναντι στη διαφοροποίηση και στην ε, διαφορετική άποψη. Είναι, πρέπει να είναι δεδομένο αυτό, διότι έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα πολύ σημαντικό φάκελο. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα στην θέση μου, επανέρχομαι ως πρόεδρος τώρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Φέντερλε είναι εδώ για να πάρει το λόγο. Όχι, δεν είναι κάποιος άλλος εδώ. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο να πει κάτι. Α, ο κύριος Τούρμες, παρακαλώ. Ναι, επειδή κάνετε σχετική αναφορά, δεν είναι για λόγους ε, κακής θέλησης που δεν συναντήσαμε την αντιπροσωπεία της Κολομβίας. Ε, Αντιλαμβάνω αυτό που λέτε, δεν, δεν ήθελα να το συναντήσω πάντως. Ένα σχόλιο μόνο για το θέμα των υλικών. Υπάρχει ένας περιορισμός. Υπάρχει όμως και μια απάντηση στον περιορισμό αυτόν. Μια εταιρεία που είναι στην πρώτη γραμμή για την αιωλική ενέργεια, η Ίνερκομ, σε λίγα χρόνια μέσω της καινοτομίας μπόρεσε να αντικαταστήσει όλο το κρίσιμο υλικό στις τουρμπίνες από μη κρίσιμο υλικό. Ε, και το, η άλλη πληροφορία που έλαβα ε, σε ό,τι αφορά τις μπαταρίες γίνονται πολλές συζητήσεις για το κοβάλτιο και στο, για το Κονγκό. Ε, το κοβάλτιο είναι υποπροϊόν χαλκού. Όπου υπάρχουν λοιπόν ορυχεία χαλκού προκύπτει και κοβάλτιο. Ε, το θέμα είναι πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια πολιτική όπου θα ανοίξουν κάποια ορυχεία στην Ευρώπη, όπως αυτό που κάνει η Σουηδία τώρα. Και είναι σημαντικό να συνδέσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες για τις βιώσιμες πηγές των ορυκτών. Ε, γίνεται δουλειά στην της Grow Επ' αυτού δεν είναι ασπρομαύρο το ζήτημα. Ε, υπάρχει ένα θέμα βεβαίως και μπορούμε όμως να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Αμπρέου Μαρκές έχει τον λόγο. Α, όχι. Όχι, εντάξει. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Προχωράμε τώρα στο EDITP. Η κυρία Κροστέτ. Επιτέλους. Oui, euh, Λυπάμαι που είμαστε τόσο λίγοι. Τουλάχιστον θα κάνω αυτή τη σύνοψη. Ήδη είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους για το πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στην άμυνα στις 15 Μαρτίου και στις 10 Απριλίου στο δεύτερο τριμερή διάλογο. Δυστυχώ, καθώ ε, δεν είχαμε συνεδρίαση της η Βουλγαρική Προεδρία, δεν έχει εντολή. Έτσι λοιπόν, δεν μπορέσαμε να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο. Απλώ αυτό μα επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξηγήσουμε εκ νέου τις θέσεις μα. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσει πρέπει να επιτεχηθούν αν θέλουμε μια ταχεία συμφωνία και είναι και πήγον σήμερα να έχουμε αυτή τη συμφωνία το συντομότερο. Συνεχίσαμε να υπερασπίσουμε την εντολή του Κοινοβουλίου με τους δύο συναδέλφους εισηγητέ από την Επιτροπή Προπολογισμού, τον κύριο Στέμπαν Γκονσαλέν Πόνς και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Πάσκου. Με τους δύο συναδέλφους πρέπει να πω ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία. Πολλά πολιτικά θέματα συζητήθηκαν και δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη. προπολογισμό ε, δεν υπάρχει πρόοδο, ήδη το ανέφερα χτε ε, στον Επίτροπο Κατάινεν, το ξανανέφερα σήμερα στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Περιμένουμε μια πρόταση τη Κομισιόν για να αποφύγουμε την ε, χρησιμοποίηση κονδυλίων από φυστάμενα προγράμματα. Αυτό συζητείται μάλιστα εδώ αυτή την εβδομάδα. Στη συνέχεια για τι μη πλέξιμες πράξεις. Μπορούσαμε να προτείνουμε μια συμβαστική εκδοχή. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία για ένα κείμενο που να αναφέρει ότι αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούν όπλα ή ε, κάποια ε, προϊόντα που έχουν απαγορευτεί από το Διεθνές Δίκαιο. Περιμένουμε την απάντηση του Συμβουλίου για τις επιλέξιμες οντότυπες. Υπενθύμησα την αγκαιότητα να πλαισιώσουμε καλύτερα την εξαίρεση που αφορά τι επιχειρήσει που ελέγχονται από τρίτε χώρε. Περιμένουμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι είναι εντελώς απαραίτητο, καθώς ε, μιλάμε για εξοπλιστικές βιομηχανίες, επομένως πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα για να γίνει σεβαστή η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Υπάρχει και μία κορεπέρ που θα συνεδριάσει αύριο, ελπίζω να συμμεθεί κάποια πρόοδο. Για το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητείται ένα συμβιβασμό για να μα επιτρέψει να αιτιολογήσουμε την προσφυγή σε εκτελεστικέ πράξει. Ε, το Κοινοβούλιο ε, ζητούσε καταξιοδότηση πράξης. Φυσικά θα πρέπει να υπερασπίσουμε τα προνόμια του Κοινοβουλίου και στον κανονισμό να διευκρινίσουμε τις κατηγορίες των σχεδίων τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Μόνο έτσι, από αυτές τις προϋποθέσεις, το Κοινοβούλιο θα μπορεί να δεχτεί την προσφυγή σε εκτελεστικές πράξεις που παίρνει λιγότερο χρόνο και μας επιτρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα για τον αριθμό των κρατών ε, μελών που απαιτούνται για τις εμπλεξιμότητες. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο περισπίσαμε το ελάχιστο των τριών επιχειρήσεων που να προέρχονται από τρία κράτη-μέλη για να συσταθεί μία σύμπραξη αντί για δύο που προτείνονται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Συζητήσαμε τη δυνατότητα να ε, υπάρξει ένα μπόνους, παραδείγματος χάρη, ε, σε ένα πρόγραμμα όπου θα συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ακόμη υποσυζήτηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δομή του μπόνους. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι αρκετά κοντά σε αυτή του Συμβουλίου. Θέλουμε να αποφεληθούν από τον σε τα σχέδια που, ε, όπου εντάσσονται οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις ή ενδιάμεσες επιχειρήσεις και θα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίσουμε ε, τους ε, τρόπους ε, χορήγησης αυτού του μπόνους τουλάχιστον για φτάσουμε σε μια συμφωνία ώστε τα ζητήματα που είναι ακόμα κρεμή και είναι πολύ σημαντικά. Ο επόμενος τριμής διάλογος είναι την επόμενη εβδομάδα, 3 Μαΐου. Κανονικά είχε προβλεφθεί στις 3 Μαΐου μια τελική συμφωνία. Φοβάμαι ότι θα χρειαστούμε ακόμη και ένα τριμήρ διάλογο μέχρι τα τέλη Μαΐου γιατί θεωρητικά θα πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο στο τέλη Μαΐου, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε το θέμα αυτό υπό Βουλγαρικής Προεδρίας και πρέπει να υπάρχει εγγραφή στον προπολογισμό, γιατί αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνος θα πρέπει να τεθεί σε από τον Ιανουάριο του 2019. Θα πρέπει επομένως να μπει στην επόμενη δημοσιονομική συζήτηση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Όμως φυσικά περιμένουμε να κάνει και το Συμβούλιο προσπάθειες από την πλευρά του. Το Κοινοβούλιο έχει θέσει κάποιους στόχους, έχουμε πει τι θέλουμε. Είπα και στον Αντιπρόεδρο Κατάινεν, σε μια διαπραγμάτευση είμαστε δύο που διαπραγματευόμαστε. Δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο από το Κοινοβούλιο να κάνει προσπάθειες και όχι από το Συμβούλιο. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε και ελπίζω να ολοκληρώσουμε καλώ αυτές τις διαπραγματεύσεις και να ξέρετε ότι τρεις εισηγητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε πραγματικά στο ίδιο μήκος και πολύ αλληλέγγυοι υπερασπιζόμαστε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη βοήθειά της, ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ. Θα τα μεταφέρουμε αυτά στον κύριο Βάρκ και στον κύριο Μπούζεκ και ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την, ε, το πόσο αποτελεσματική είναι η γραμματεία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, τα διάφορα. Να σας ενημερώσω ότι 17 Μαΐου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για την επιστήμη και την καινοτομία, ενίσχυση της διεθνής συνεργασίας στο πλαίσιο του ενάτου προγράμματος πλαισίου. Θα οργανωθεί σε συνεργασία με το πάνελ ΣΤΟΑ. Ε, και την STS που είναι το ε, αντίστοιχο της Ιαπωνέζικης ΣΤΟΑ. Και προχωρώ στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διάταξης. Η επόμενη συνάντησή μας ε, θα είναι στις 16 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 2.30 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Και 17 Μαΐου, 9 με το 10.30 και πάλι από τις 3 το απόγευμα έως τις 6.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λήξη της συνεδρίασης.